Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Euh, Έχουμε πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη, γι' αυτό καλό θα ήταν να μην καθυστερούμε άλλο. Και το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά πιστικό για σήμερα το απόγευμα. Καταρχήν, έχετε κανένα πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη? Όχι, οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αμετάβλητη. Επίσης, ε, ε, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο web streaming και έχουμε και διερμηνία σε 16 γλώσσες. Και να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία τους διερμηνείς από τώρα. Για τα πρακτικά τώρα. Έχετε λάβει διάφορα πρακτικά από τις συνεδριά της 8 Σεπτεμβρίου και 12 και 13 Οκτωβρίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Και να περάσουμε στο κυρίως θέμα της απογευματινής μας ημέρησης διάταξης, τη δημόσια ακρόαση με θέμα μια γεωργία φιδωλή ως προς τους πόρους και καινοτόμο βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Θα χωρίσουμε τη δημόσια ακρόαση σε δύο τμήματα, γι' αυτό και θα είμαι κάπως αυστηρός ε, στη χορήγηση του χρόνου. Το πρώτο τμήμα θα μιλήσουμε για τις βέλτιστες πρακτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ακούσουμε τον κύριο Πρωταμπέλα Γκλατμπέλντερ, τον πρόεδρο της πλατφόρμας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Ουγγαρία, κατόπιν τον καθηγητή Φιλίπ Μπαρέ του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβά στο Βέλγιο και τρίτον τον δόκτωρα Κέβιν Μορέλ από το Πανεπιστήμιο Σακλέ της Γαλλίας. Δέκα λεπτά θα έχει ο κάθε καλεσμένος. Θα ακολουθήσει ένας γύρος ερώτα απαντήσεων και ελπίζω στο μεταξύ να καταφτάσουν και άλλα μέλη της Επιτροπής για να λάβουν μέρος στη συζήτηση και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης στο οποίο θα μιλήσουμε για τις βέλτιστες πρακτικές στον κόσμο με δύο ομιλίες του καθηγητού Σίναν Χάρπας από την Οργάνωση για τη Γεωργική Έρευνα στο Κέντρο Βολκάνη του Ισραήλ και του καθηγητού Πάτρικ Worms από το Παγκόσμιο Κέντρο Αγροδασοκομείας του Βελγίου. Δέκα λεπτά θα έχουν και οι καλεσμένοι του δεύτερου γύρου και κατόπιν θα γίνει συζήτηση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις λοιπόν, θα περάσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στην πρώτη παρουσίαση του κυρίου Μπέλα Γκλάτφελντερ από την Ουγγαρία. Έχετε 10 λεπτά και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την τήρηση του χρόνου. Ευχαριστώ. Ε, ήμουν και εγώ μέλος της Επιτροπής ε, για πολλά χρόνια, δέκα χρόνια και χαίρομαι που ξαναβλέπω οικία πρόσωπα, φίλους και γνωστούς. Με προειδοποίησαν όμως ότι καλό θα ήταν να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα συνεχίσω λοιπόν στα Ουγγρικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα σας μιλήσω για, μεταξύ για τη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειών σε ποιε εξοικονομήσει διοξιδίου του άνθρακο και σε ποιε εξοικονομήσει ενεργεία μπορούμε να καταλήξουμε με τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειών στην γεωργία. Θα ενθυμίσετε ίσω το γράφημα που σας δείχνω στον ε, πίνακα που ε, είχα φτιάξει όταν ήμουν εισηγητή στην Επιτροπή Γεωργίας και είχαμε πει ότι μέχρι το 2050 θέλαμε να μειώσουμε κατά 80% το διοξίδιο του άνθρακος. Και αυτό αποτελούσε μάλιστα και οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε αυτόν τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούσαμε επίσης για το γεγονός ότι έχουμε κάποιες περιορισμένες δυνατότητες στην ε, Γεωργία διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι δεν μπορεί να μειωθεί η εκπομπή διοξιδίων του άνθρακος πάνω από 45%. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίξει ωστόσο σημαντικό ρόλο και η μεταποίηση τροφίμων, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε τρόφιμα. Θεωρώ ότι η παραγωγή τροφίμων λοιπόν έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο από, άλλη, από άλλους κλάδους της γεωργίας. Τις μεγαλύτερες εξοικονομήσεις μπορούμε να τις επιτύχουμε στην Ήπεθρο και οι Ευρωπαίοι γεωργοί, οι Ευρωπαίοι αγρότες, επενδύουν σημαντικά στις ανανεώσιμες ενέργειες. Μεταξύ 2009 και 2013 οι Γερμανοί οι γεωργοί επένδυσαν 19 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανανεώσιμες ενέργειες. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, 40% από την παγκόσμια κατανάλωση ε, καυσίμου γίνεται στην γεωργία και υπάρχουν εδώ διάφορες δυνατότητες που, ε, και μέθοδοι που μπορούν να επιτρέψουν και άλλες εξοικονομήσεις. Η γεωργία μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο τα βιολογικά καύσιμα. Όμως τα σημερινά ε, φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται δεν δίνουν αρκετά κίνητρα. Κάτι άλλο που καταναλώνει πολύ ενέργεια είναι η άρδευση. Αν όμως δεν αρδεύουμε, τότε θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια για άλλες δραστηριότητες της γεωργίας. Δυστυχώς, ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες δεν είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο που να προσφέρουν κίνητρα για μια βελτίωση της ε, χρήσης ενέργειας στην άρδευση ανά εκτάριο μπορεί ένας γεωργός στην Ουγγαρία να εξοικονομήσει 50 λίτρα καυσίμου δίζελ εάν χρησιμοποιήσει, αν επιλέξει ε, καινοτόμες μεθόδους άρδευσης. Σε ό,τι αφορά την ξύρανση, στην ε, Ουγγαρία υπάρχουν δύο μεγάλες εγκαταστάσεις αποξύρανσης, οι οποίες ε, κινούνται με βιοθερμική ενέργεια. Οι υπόλοιπε ε, αντρούν την ενέργεια από παραδοσιακές πηγές. Στην ξύρανση, από την ξύρανση μάλλον, προκύπτουν πολλά υποπροϊόντα, τα οποία μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Η κτηνοτροφία επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Το βιολογικό αέριο μειώνει βεβαίως την ε, ε, χρήση ενέργειας στην γεωργία, αλλά από την άλλη μεριά αποδίδει και αυτό στην ατμόσφαιρα ε, οξύδια του άνθρακα. Δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκοί μάλλον ή εθνικοί νόμοι που να ε, προσφέρουν κίνητρα για τη χρήση σε μεγαλύτερη κλίμακα του βιολογικού αερίου. Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις οι οποίες καταναλώνουν και ηλεκτρικό ρεύμα αλλά επίσης παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα και θερμότητα, θερμική ενέργεια και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να επιτρέψουν στον αγρότη να εξοικονομεί σημαντικά ποσά. Επίσης, στην οικοδομή έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν, ε, κατασκευάζονται πλέον οι στέγες των κτηρίων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν και στα γεωργικά κίνητα να ε, εγκαθίστανται ε, ηλιακές εγκαταστάσεις. Βλέπετε εδώ επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γεωργού, ο οποίος καλλιεργεί πάπρικα στην Ουγγαρία και θερμένη τις εγκαταστάσεις του με βιοθερμική ενέργεια. Στην Ουγγαρία η βιοθερμική ενέργεια παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ιδίως στην παραγωγή οπροκυπευτικών. Ασφαλώς δεν πρόκειται μόνο για βιοθερμική ενέργεια. Με τα διάφορα παραγόμενα υποπροϊόντα της γεωργίας, αυτά επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή θερμότητας, τα απόβλητα της γεωργίας μπορούν και αυτά δηλαδή να καίονται για να προσφέρουν ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ε, χρήση, τη μεταποίηση τροφίμων, παροιμήν χρησιμοποιούνται διαδικασίες χαμηλής ε, ε, θερμοκρασίας, χαμηλής θερμότητας, αντίθετα από τη χαλιβουργία για παράδειγμα, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ανανεώσιμες ενέργειες λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται σε εμά όμως, δηλαδή στην μεταποίηση ε, γεωργικών προϊόντων για την ε, παραγωγή τροφίμων, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλότερε θερμοκρασίε και επίση παράγονται, όπω είπα, υποπροϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ε, βλέπετε εδώ μία, είδατε μάλλον, μία μεγάλη εγκατάσταση που περιλαμβάνει ορνηθοτροφείο και ε, εκεί προβαίνουν στην μεταποίηση του κρέατος πουλερικών και χρησιμοποιούνται τα απόβλητα για την θέρμανση. και μάλιστα μέχρι, ε, φτάνουν μέχρι να παράγουν και 4 ΜΒ την ώρα. Επίσης ε, κατά την μεταποίηση ελαιοδών σπόρων. Εκεί χρησιμοποιούνται τα, χρησιμοποιούνται ο φλοιός των σπόρων, των ιδιόσπορων δηλαδή, για την ε, παραγωγή ενέργειας και μάλιστα η, παραγωγή ενέργειας υπερβαίνει την κατανάλωση ε, που ε, απαιτείται για την εγκατάσταση, άρα περισσεύει. Αλλού χρησιμοποιούνται τα πριονίδια. Σε μια μικρή πόλη στην Ουγγαρία παράγεται, παράγεται συγκεντρω, ε, συγκεντρωμένος ε, τοματοπολτός και εκεί χρησιμοποιούν και τον φύλλο της τομάτας και τους σπόρους για την παραγωγή ενέργειας. Δηλαδή τα καίνε, ενώ παλιά απλώς τα πετούσαν. Χρησιμοποιούνται λοιπόν τώρα και αυτά. Στην Ουγγαρία υπάρχει και μια ε, εγκατάσταση παραγωγής ισογλυκόζης στην οποία χρησιμοποιούνται οι φλοί των ιδιόσπορων και ο σανός και χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας με αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση. Και μάλιστα ε, η παραγωγή του φτάνει για να ηλεκτροδοτήσει μια πόλη 120.000 κατοίκων για ένα χρόνο. προχωρούν σε επενδύσεις οι γεωργοί και με κίνητρα που τους παρέχονται και σωστό είναι να χρηματοδοτούνται επενδύσεις οι οποίες δεν αυξάνουν την ε, εκπομπή του διοξιδίων του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους έργα που χρησιμοποιούν παραδοσιακές πηγές ενέργειας ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ουγγαρία έχω επισκεφθεί εγκαταστάσεις που θερμαίνουν κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις με ορυκτά καύσιμα ενώ στις περιοχές αυτές υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο το βιολογικό αέριο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, λοιπόν, όπου μπορούν να βοηθήσουν και οι ευρωπαϊκοί ε, νόμοι, ενώ στην πραγματικότητα μέχρι τώρα συχνά παρεμβάλλουν εμπόδια. Έχουμε λοιπόν μεγάλο δυναμικό και αυτό μπορεί να μεγαλώσει ακόμη. Βλέπετε στην εικόνα που δείχνω τώρα, με το γκούλα, βλέπετε το ουγγρικό ε, παραδοσιακό φαγητό, το οποίο και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν τέλει για την παραγωγή ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Σας ευχαριστούμε κύριε Γκλάτπλαντερ και συγχαρητήρια για την ε, αυστηρή χρήση του χρόνου. Δείξτε την ίδια συνέπεια και ακρίβεια όταν ήσασταν μέλος της Επιτροπής. Και τώρα ο κύριος Μπαρέ από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβά. Επίσης για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στόχος μου σήμερα είναι να σας μιλήσω για τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια αποδοτική στη χρήση των πόρων γεωργία και να σας πείσω ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτή η πρωτοβουλία αφορά όχι μόνο τη γεωργία αλλά και το επιστηστικό σύστημα γιατί δεν μας παίρνει πια να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να μειώσουμε τις επιπτώσεις της γεωργίας και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τις πρακτικές ε, της γεωργικές. Θα πρέπει όμως να δώσουμε καινούργια κίνητρα και τα κίνητρα αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από πολιτικό επίπεδο, είτε από, από τους καταναλωτές, είτε από το συνδυασμό και των δύο. Οπότε το, οι επιπτώσεις και οι αλλαγές επεκτείνονται στο σε ολόκληρο το πιστιστικό σύστημα. Και μετά την ε, επανάσταση της παραγωγικότητας του 20ου αιώνα και με την, μετά την Πράσινη Επανάσταση, σήμερα διαπιστώνουμε την ανάγκη να αποκτήσουμε μια νέα ατζέντα για τη Γεωργία. Και ο Ολιβιέντε Κουτέρο, ειδικό ε, εισηγητή των Ηνωμένων ε, στην έκθεση του 2010, υπενθυμίζει ότι οι τρει βασικέ προκλήσει τη γεωργία σήμερα είναι το δικαίωμα στην σύντηση, δηλαδή ο κόσμο θα πρέπει να μπορεί να ε, λαμβάνει το τρόφιμα που χρειάζεται. Δεύτερον, ισότητα, να μειωθούν οι ανισορροπίες και οι ανισότητες μεταξύ των γεωργών, κυρίως μεταξύ Βορρά και Νότου. Και οι γεωργοί του Νότου είναι από τις φτωχότερες ομάδες του πλανήτη και επίσης ε, βιωσιμότητα, αηφορία. Αυτή είναι η τρίτη πρόκληση της γεωργίας. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο γεωργίας που να το χρησιμοποιούμε στα διενεκές, δηλαδή να μην ε, υπονομεύσουμε την μελλοντική γεωργία με τις σημερινές πρακτικές. Οπότε δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην παραγωγή αλλά και στο γεωργικό εισόδημα και στη βιωσιμότητα. Επίσης να δούμε τις προσδόκητες επιπτώσεις γεωργίας και να αλλάξουμε τις επιπτώσεις, κυρίως τις επιπτώσεις γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές. Και επίση θα πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο τη εντατικοποίηση. Μέχρι την αρχή του 21ου αιώνα η εντατικοποίηση οδηγούσε σε αύξηση τη απόδοσης και δεν είχε αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Στον 21ο αιώνα όμως είχαμε τριπλασιασμό των αποδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός όμως ο τριπλασιασμός της απόδοσης είχε και κάποιες ε, πολύ επιζήμιες εξωτερικές ε, συνέπειες ε, στη ρήπαση του εδάφους, των αποδοσεων σε παγκοσμιο επιπεδο αυτος ομως ο τριπλασιασμος της αποδοσης εχει και επηρέασε αρνητικά και το περιβάλλον. Και πάλι, γι' αυτό δεν μπορούμε στον 21ο αιώνα να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Και μάλιστα Έχουμε εδώ στον κύκλο το στόχο για το 2050. με πορτοκαλί χρώμα έχουμε τα κέρδη από την παραγωγικότητα, διπλασιασμό των κερδών και σε πράσινο τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σε ό,τι φορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας. Έχουμε λοιπόν διπλούς στόχους. Θα πρέπει αφενός να αυξήσουμε την παραγωγή και αφετέρου να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που αν συνεχίσουμε στο business as usual σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ε, δεν δεν, έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πια κάτι τέτοιο. Α, αριστερά έχουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και δεξιά τις επιπτώσεις ό,τι αφορά τις αζωτούχες ενώσεις, τις επιπτώσεις των περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τις επιπτώσεις της γεωργίας χωρίς ταυτόχρονα να μειώσουμε και την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα. Από τεχνική άποψη είναι δύσκολη υλοποίηση αυτού του στόχου. Ε, μεταβατικά τουλάχιστον θα πρέπει να αποδεχθούμε και μία μείωση της αποδοτικότητας, κάτι που δεν είναι ασυμβίβαστο με τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι η ένδυα στον κόσμο και όχι η παραγωγή. Ε, επίσης, ένα θέμα των παραγωγών παγκοσμίω είναι ακόμη στην αφετηρία και αυτή δεν χρειάζεται να περάσουν στη φάση της, ε, της γεωργίας με αρνητικές συνέπειες, θα μπορούσαν να περάσουν κατευθείαν σε μια γεωργία, τη βιολογική για παράδειγμα, που δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο στόχος και της αγροοικολογίας. Επίσης, ε, δεν είναι απαραίτητο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Βλέπουμε στην πρώτη γραμμή την αύξηση τη παραγωγικότητα ε, και την επίπτωση στα τρόφιμα. Στα, ε, στην κόκκινη γραμμή έχουμε τη δημογραφική αύξηση. Σε αρχέ τη δεκαετία του 60 η παραγωγικότητα ανακάτοικο αυξάνεται. Έχουμε όμω 830 εκατομμύρια συνανθρώπου μα που υποφέρουν από υποσυτισμό και πείνα. Και έχουμε πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα αυτό και την έκθεση του Λιβέντε Σκουτέρ οι προκλήσει είναι πολύ περίπλοκε. δεν αφορούν μόνο την παραγωγικότητα, αφορούν κυρίω την εξάλληψη τη φτώχεια και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Τι γίνεται με την αγροοικολογία, γιατί πολύ την αναφέρουμε. Είναι θέμα αρχή περισσότερο. Μιλούμε για αγροοικολογικέ πρακτικέ που έχουν κάποιο ενδιαφέρον, αλλά η αγροοικολογία από πανεπιστημιακή άποψη στηρίχθηκε σε κάποιες αρχές. Στις αρχές της οικολογίας, φιδωλή χρήση των πόρων για παράδειγμα, κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα βιοπικιλότητα, χρήση της ανακύκλωσης, ε, ενδιαφέρον για το έδαφος και κάποιες παιδαγωγικές αρχές, οικολογικό σχεδιασμός, οικολογική καινοτομία, συμμετοχή και κάποιες κοινωνικο-οικονομικές αρχές, ε, συνεργασία, ε, fair trade, δίκαιες τιμές, δίκαιο εμπόριο και σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού. Επίσης, έχουμε τη συστημική διαίρεση που σημαίνει ε, μια διαίρεση που εδράζεται στις αλληλεπιδράσεις και έχουμε πολλά σημεία εξόδου και όχι μόνο την παραγωγικότητα και αναζητούμε τις καλύτερες ε, συμβαστικές λύσεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα και δεν είμαι ο μόνος ε, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μία μετάβαση. Θα πρέπει να αφήσουμε ένα σύστημα που έχει ένα και μοναδικό στόχο την ε, βελτίωση της παραγωγικότητας και το τη διαφύλαξη του εισοδήματος των μεγαλύτερων ε, γεωργών, να μεταβούμε προς ένα σύστημα πολυμορφίας και πολυλειτουργικότητας που θα έχει output και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Επίσης αυτή η μετάβαση θα πρέπει να δράζεται σε μια συστημική προσέγγιση και να μην είναι ένα άθροισμα καλών και, ε, πρακτικών και παραδειγμάτων. Η συστημική προσέγγιση θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο ε, του προβληματισμού μας. Και εδώ γιατί. Έχουμε μια μελέτη που έγινε στο Βέλγιο με διαφορετικά είδη παραγωγής, γάλακτο παραγωγής. Μερικά στηρίζονται στα, στα λιβάδια και άλλα στη χρήση αραβόσιτος ζωοτροφής. Και το σύστημα που στηρίζεται σε τέτοιες ροές είναι το πιο θετικό από οικονομική άποψη. Και τα το, που στηρίζονται σε λιβάδια με πράσινο δεν είναι πολύ αρνητικά από οικονομική άποψη και οικολογικά είναι πολύ πιο επωφελή. Οπότε η επιλογή μας ε, θα είναι αμυγός οικονομική ή θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος. Επίσης έχουμε μερικούς ε, γεωργούς που βρίσκονται στο κόκκινο, που δεν τα βγάζουν πέρα. Οπότε το θέμα είναι τι ε, κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν την πιο ενδιαφέρουσα κατεύθυνση από οικονομική άποψη ή την πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση από οικολογική άποψη. Και αυτή τη μετάβαση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη τους δύο άξονες, τον περιβαλλοντικό άξονα με χ και τον κοινωνικο-οικονομικό άξονα που αναφέρεται εδώ με y με y. Ε. Και στην κοινωνικονομική διάσταση έχουμε και το θέμα της απασχόλησης, γιατί από τις βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα στη Γεωργία στην Ευρώπη είναι να εξασφαλίσει ανάπτυξη της υπαίθρου και θέση εργασίας στην υπαίθρο. Οπότε οι διαστάσεις αυτές ε, της απασχόλησης, η κοινωνικο-οικονομική, ε, μας ενδιαφέρουν κυρίως στους καταναλωτές και για τη δημόσια πολιτική, ενώ η περιβαλλοντική διάσταση βρίσκεται κυρίως στα χέρια των γεωργών. Τώρα, στο σύστημα αυτό η θέση των διαφόρων ε, συστημάτων εξαρτάται από τις ε, δημόσιες, πολιτικές. Τι δημόσιε πολιτικέ και κυρίω ε, την πολιτική των τιμών. Αν αλλάξουμε τι τιμέ των βιολογικών προϊόντων, αλλάζουν οι θέσει στο σύστημα. Οπότε θα πρέπει να επιλεγούν διαφορετικέ συμβαστικέ λύσει κάθε φορά. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε από μία σκέψη που εδράζεται αποκλειστικά και μόνο στον γεωργό και στην παραγωγή και να μεταβούμε προ μια σκεψη που λαμβανει υποψη ολοκληρη την αλυσιδα τη αξία απο το γεωργο προσέγγιση. Τώρα, σε αυτό το σύστημα μπορούμε να επηρεάσουμε τις τιμές. Βέβαια, εκεί οι μεγάλες αλυσίδες διανομής επηρεάζουν ε, τον καθορισμό τους. Ή μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο περίπλοκο το σύστημα και να πούμε ότι το, ούτως ή το επιστηστικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο και μάλιστα σας δείχνω αυτή την εικόνα μιας βελγικής εταιρείας ε, με συνεργασία του συναδέλφου Ρίκ Ματέης από το Πανεπιστήμιο του Σιλουβά. Εμείς βρισκόμαστε εκεί πάνω, στο πάνω μέρος του της απεικόνησης αυτής. Και οι πολιτικοί θύνοντες ε, ε, πειράζουν και τους γεωργούς και τους καταναλωτές και τη σχέση γεωργών και καταναλωτών με τις αποφάσεις τους. Οπότε, ως πανεπιστημιακός, ε, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται μια δημόσια πολιτική και μια δημόσια δράση, γιατί θεωρώ ότι η βιωσιμότητα της γεωργίας μας και μιας γεωργίας αποδοτικής στους πόρους απαιτεί συμβαστικέ λύσει, γιατί η περισσότερη βιωσιμότητα προποθέτει ελαφρά μεν, αλλά μείωση δε της παραγωγικότητας. Οπότε, όταν έχουμε μείωση τη παραγωγικότητα, θα αλλάξει και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Θα πρέπει να είναι καταρχήν ο καταναλωτή έτοιμο να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή για το τρόφιμα, για τη διατροφή του και σε παγκόσμια κλίμακα θα γίνουν κάποιε αλλαγέ ε, σε ό,τι αφορά τι συνήθειε τι διατροφικέ ε, ίσως από τη θετική στη ζωική περισσότερο ε, κατανάλωση από περισσότερο ζωικών προϊόντων. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη ισοτιμία και δικαιοσύνη μεταξύ των, των γεωργών. Ε, δεν θα πρέπει να είναι ο στόχος ε, μόνο η μεγέθυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γιατί με ένα τέτοιο μοντέλο, ξεχάστε τους γεωργούς, έχουμε απλώς ε, μεγαλογεωκτήμονες διαχειριστές απλώς τεράστιων γεωργικών εκτάσεων. Δεν θα είναι όμως πραγματικοί γεωργοί. Και τώρα πώς θα έχουμε αύξηση της ισότητας, της ισοτιμίας, θέλουμε αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων εντός των ε, επιστηστικών συστημάτων. Και αυτή η αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων δεν μπορεί να γίνεται απλώς με τα λόγια. Θα πρέπει να προηγηθεί ένας εντοπισμός και εξάλληψη των παραγόντων ε, ε, του εγκλωβισμού σε συγκεκριμένους κανόνες και από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως συμβαίνει σήμερα. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ότι ε, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μιας γεωργίας που θα είναι αποδοτική ως προς τους πόρους θα πρέπει να εντοπίσει και να ξεπεράσει αυτά τα κολλήματα και να δημιουργήσει περισσότερες ικανότητες, να προασπίσει κάποιες θετικές πρωτοβουλίες. Θα δούμε τέτοια παραδείγματα σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να προτείνει τα μοντέλα που θα είναι κατάλληλα στους σύγχρονους, για τους σύγχρονους γεωργούς, γιατί η σύγχρονη γεωργία θα είναι οι φορείς της μετάβασης και επίση χρειάζεται μια συνέπεια στι δράσει, στι ενέργειε. Δηλαδή να μην ζητούμε από του γεωργού να κάνουν κάτι και με το επιστημιστικό σύστημα να του βάζουμε τροχοπέδι σε αυτέ τι προσπάθειες. Και αυτό είναι το θέμα τη συνέπειας στη δράση. Και ποιο είναι το βασικό μου μήνυμα. Για να αλλάξουμε τις επιπτώσεις θα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα τις πρακτικές. Χρειάζεται τεχνολογική επανάσταση, αλλά χρειαζόμαστε και νέα κίνητρα για τους γεωργούς. Αυτή θα είναι η κοινωνικο-οικονομική επανάσταση που θα πρέπει να συνοδεύει την τεχνολογική. Επίσης θα πρέπει να τροποποιήσουμε τα επισητιστικά συστήματα και γι' αυτό χρειάζεται και ένα πολιτικό όραμα και πολιτικές αποφάσεις που θα στηρίξουν αυτές τις μεταβάσεις. Οπότε η μετάβαση δεν είναι μόνο ένα σύνθημα, ένα σλόγγαν. Ε, προποθέτει σημαντική έρευνα και πολλοί ερευνητέ ασχολούνται με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρέ, για αυτές τις πλούσιες και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και θα δώσω αμέσω ε, το λόγο στον ε, κύριο Κεβιν Μορέλ ε, για την τρίτη παρέμβαση για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εγώ θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα Έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένες μελέτες εκμεταλλεύσεων στη Βόρεια Γαλλία και η καινοτομία η οικολογική μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερους πόρους αλλά να έχουμε και ψηλό επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας και όπως ξέρετε αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και φυσικά η καινοτομία γίνεται σε επίπεδο εκμετάλλευση αλλά και σε ευρύτερη συλλογική δυναμική. Εγώ εργάζομαι σε πολύ συγκεκριμένα συστήματα που τα λέμε μικροεκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη Γαλλία και έχουν αυξανόμενη επιτυχία. Έχουμε πάρα πολύ μικρές ε, εκμεταλλεύσεις ε, που παράγουν λαχανικά και έχουμε νέους αγρότες που δεν προέρχονται από αγροτικό περιβάλλον, συχνά έχουν υψηλό εκπαιδευτικό μορφωτικό επίπεδο και ασχολούνται με τη γεωργία γιατί θεωρούν ότι έτσι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι νέοι γεωργοί φτάνουν στις εκμεταλλεύσεις και δεν θέλουν να εγκατασταθούν σε πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αντιθέτως επιλέγουν πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις με μεγάλη ποικιλομορφία οικολογικών πρακτικών. Παραδείγματος χάρη εδώ ε, έχουμε κάτω από 1,5 εκτάριο ανά άτομο με ανθρώπους. Εδώ βλέπετε το χάρη σε ένα τετραγωνικό μέτρο μπορεί να έχουμε μια σαλάτα παραβίκια και από κάτω καρότα και δίνεται και μεγάλη σημασία στους ε, οικοτόπους επίσης. Ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν και τοπικές δυναμικές οι άνθρωποι αυτοί συνεργάζονται με τα χωριά τριγύρω, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη στην υπεθρο, Μπορεί να σας ε, φαίνονται ουτοπικά όλα αυτά, όμως εμείς προσπαθήσαμε να δούμε στην έρευνά μας αν αυτές οι πρακτικές μπορούσαν να συμβάλλουν και να οδηγηθούν σε οικονομική βιωσιμότητα. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης σε 20 μικροεκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Γαλλία. Εδώ Προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τρία συστήματα. Στον τρίτο πίνακα, δεξιά, ε, βλέπετε ε, ουσιαστικά την ε, ε, κυπουρική για την αγορά και εδώ έχουμε ένα τρακτέρ για να κάνουμε τις περισσότερες δραστηριότητες, την άρρωση του εδάφους και τις βαριές δουλειές και χρησιμοποιούνται και ε, λιπάσματα και φυτογενομικά προϊόντα. Δεξιά εδώ έχουμε τα άλλα σενάρια δίπλα, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, μικρότερες εκτάσεις και όπως σας είπα χρησιμοποιούνται πράσινα λιπάσματα και έχουμε και το πρώτο σενάριο και δεν υπάρχει καθόλου μηχανοκίνητη μηχάνηση της γεωργίας και ε, εδώ υπάρχει ε, ε, μια ουσιαστικά πολύ έντονη χειρονακτική εργασία και υπάρχει μια ελαφριά δουλειά στο έδαφος. Ε, βλέπετε εδώ τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στα δύο πρώτα συστήματα έχουμε τις μικροεκμεταλλεύσεις και αν το συγκρίνουμε με το πιο κλασικό σύστημα αυτά, καταναλώνουν ε, λιγότερη ενέργεια γιατί έχουμε μικρότερη εκμηχάνηση και επίσης ε, καθώς δεν υπάρχει άρρωση του εδάφους, δεν υπάρχει και διάβρωση του εδάφους και καθώς χρησιμοποιούν οικολογικές πλακτικές επίπεδο εκμετάλλευσης, ε, ε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγα λοιπάσματα και φυτογενομικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας και όσο αφορά την ε, βιοπικιλότητα ε, βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτό και αν δούμε και την οικονομική βιωσιμότητα, βασιζόμαστε εδώ σε πραγματικές εκμεταλλεύσεις, αλλά καθώς είναι πολύ λίγες και είναι πρωτοπόρες έχω βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα για να διερευνήσω με δημιουργία μοντέλων κάποια σενάρια. Για κάθε εκμετάλλευση εδώ έχω δοκιμάσει χίλια σενάρια και βλέπετε ότι κατά μέσο όρο η πρώτη ε, εκμετάλλευση, η μικροεκμετάλλευση παράγει περισσότερο ανά μονάδα επιφάνειας. Ε, έτσι λοιπόν δεν έχουμε εδώ απόδοση των νεκταρίου αλλά σε ό,τι αφορά το εβδομαδιαίο καλάθι λαχανικών. Ένα πλήρες καλάθι λαχανικών για μία οικογένεια, για μία εβδομάδα επί 50 εβδομάδες και πόσο μπορούμε να παράγουμε, πόσα καλάθια νεκτάριο. Και βλέπετε ότι τα δύο πρώτα στήματα που είναι πολύ οικολογικά, στην πρώτη περίπτωση έχουμε περίπου 100 καλάθια, στη δεύτερη ε, περίπου 90 και ε, ε, ε, όταν πάμε στο τελευταίο είμαστε στα 25, δηλαδή έχουμε λιγότερη εκμεχάνηση και μπορούμε να αντικοποιήσουμε την καλλιέργεια. Γιατί, ε, παραδείγματο χάρη, όταν δεν έχουμε πλέον τρακτέρ μπορούμε να έχουμε πιο πυκνές καλλιέργειες και με το ανθρώπινο χέρι μπορούμε να παράγουμε περισσότερα. Και σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα βλέπετε ότι φτάνουμε σε δυνατότητες ανώτερες ε, για το σενάριο της μικροεκμετάλλευσης σε σχέση με το κλασικό σενάριο. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι έχουμε εδώ ε, μιλήσει για τις πιο μικρές επιφάνειες και βλέπουμε ότι έχουμε 3.000 τετραγωνικά μέτρα, 6.000 τετραγωνικά μέτρα ανά γεωργό, ενώ στο κλασικό έχουμε περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα και επομένως μπορεί να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας για ε, μια μικρότερη επιφάνεια. Οι γεωργοί προσπαθούν επίσης να συνεργαστούν με το οικοσύστημα, αλλά και να συνεργαστούν και με τους γειτονές τους ε, και όχι μόνο με τους ανθρώπους ε, με τους οποίους έχουν το ίδιο όραμα αλλά και με πιο συμβατικούς γεωργούς. Βλέπετε παραδείγματο χάρη εδώ μια συνεργασία μεταξύ γεωργών ε, στη, στη Βρετάνη. Έχουμε μια μικροκμετάλλευση βιολογική. Συνεργάζονται οι άνθρωποι αυτοί και με ένα γαλακτοκομείο 80 εκταρίων και με μια ζηθοποιία και ε, όσο οργανώνονται οι άνθρωποι αυτοί, ε, τελικά φαίνεται ότι είναι καλό να δουλεύει κανεί σε επίπεδο εκμετάλλευση, αλλά υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των εκμεταλλεύσεων. Γιατί κάποιε εκμεταλλεύσει ε, θα παράξουν, παραδείγματο χάρη, απόβλητα και μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν από άλλε εκμεταλλεύσει. Και καθώ συνεργάζονται λοιπόν αυτέ οι εκμεταλλεύσει, μπορούμε να κυκλώσουμε μία σειρά υλικών τοπικά και αυτό μας ε, επιτρέπει να μην ε, προσφύγουμε σε εξωτερική βοήθεια. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ ότι η μικρή εκμετάλλευση και η γεωτικομία ε, χρησιμοποιούν ένα τρακτέρ και μπορούν να περιορίσουν την ενέργεια και βλέπετε ότι οι τρεις επιχειρήσεις ε, ουσιαστικά δημιουργούν μια μηβαία σχέση για να πουλήσουν μαζί στην αγορά. Και τελικά, αν οργανωθούμε σε επίπεδο επικράτειας, μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότερους πόρους, αποδοτικότερων πόρων. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των γεωργών έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην τοπική ζωή γιατί με τη συνεργασία των γεωργών δημιουργούν ε, ε, μια ελκυστική επικράτεια είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συνεργασία του και υπάρχουν άνθρωποι που λένε Α, και εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλε δραστηριότητε, που χάρη να παράξουμε τυρί με το γάλα, και σε επίπεδο χωριού έχουν δημιουργήσει μια τέτοια δυναμική που το χάρη βλέπετε κάτω δεξιά στη φωτογραφία έχουμε ένα χωριό το οποίο ήταν υποερήμωση και υπάρχουν τώρα νέοι άνθρωποι που εγκαθίστανται και κατασκευάζουν, κατασκευάζουν τα σπίτια γιατί βλέπουν ότι αποκτά ζωή το χωριό έτσι λοιπόν έχουμε αντίκτυπο και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Δυστυχώς είναι πολύ μικρά η οθόνη και δεν βλέπουμε εδώ καλά αλλά θα σας τα πω για να με ακούσετε. Βλέπουμε εδώ ότι αυτή η συνεργασία επιτρέπει την βελτίωση της χρήσης των πόρων και όταν μιλάμε για την αποδοτικότητα των πόρων στη γεωργία, οι πολιτικές δεν πρέπει να επικεντρώνουν σε επίπεδο εκμετάλλευσης, αλλά να έχουμε μία διάσταση ε, που αφορά την επικράτεια και είναι πολύ σημαντική η διάσταση αυτή για την καινοτομία. Γιατί όταν θέλουμε να έχουμε πρακτικές που να βασίζονται στο οικοσύστημα, οι γενικές αρχές που έχουμε στο εργαστήριο δεν δουλεύουν πια. Γιατί το οικοσύστημα είναι κάτι πολύπλοκο, πρέπει να ξέρουμε το έδαφος, το κλίμα και αυτό δεν μπορούμε να το αναπαράξουμε στο εργαστήριο. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στο έδαφος και όσοι γνωρίζουν τη γη είναι η γεωργοί. Έτσι λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε επιστήμη και να έχουμε μια εταιρική σχέση μεταξύ επιστημόνων και γεωργών και συλλογικά, γιατί οι γεωργοί ε, ουσιαστικά συζητούν μεταξύ τους και τους αρέσει αυτό. Βλέπετε και την εικόνα ψηλά δεξιά. Έχουμε μία μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στη Λορένη από το Υπουργείο Γεωργίας εδώ. Ε, ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκε ένα σύνολο εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν οικολογικές πρακτικές, ε, χειρονακτικά εργαλεία που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για τη χειρονακτική εργασία και είχαμε πολύ καινοτόμα πράγματα Παραδείγματος ε, χάρη έχουμε ουσιαστικά εργονομικά σχέδια για τα εργαλεία τα οποία τώρα είναι στο διαδίκτυο και είναι ανοιχτά. Έτσι λοιπόν όπως ε, σας είπα αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε και μια τοπική δυναμική που έδωσε ανάπτυξη στην Ήπεθρο και έδωσε και ε, τη βούληση στους ανθρώπους να εγκατασταθούν στην περιοχή. Το 2000 είχαμε περίπου 8 τέτοιες εκμεταλλεύσεις και μετά, ε, μετά από 15 χρόνια φτάσαμε στις 120 και αυτό οφείλεται σε αυτή την συλλογική δυναμική. Για να συνοψίσω ό,τι αφορά τώρα τις επιπτώσεις για την κοινή αγροτική πολιτική, όπως σας είπα, οι γεωργοί, ε, καθώς έχουν μικρές επιφανίες, ε, συνήθως ε, δεν αποφελούνται τόσο από την κοινή γεωργική πολιτική, όσο οι υπόλοιποι. Παρόλα αυτά, είναι η δουλειά της πιο οικονομικά βιώσιμη γιατί ξέρουν ότι δεν θα έχουν βοήθεια από την ΚΑΠ, έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουν περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο πρώτου πυλώνα θα ήταν πιο ενδιαφέρον να δίνουμε τι ενισχύσει ε, αναγεωργό παρά αναεκτάριο, γιατί μιλάμε για ανθρώπου που έχουν πολύ μικρή επιφάνεια γη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, θα ήταν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουμε και να στηρίξουμε τη συλλογική καινοτομία, γιατί αυτή η συλλογική δυναμική μπορεί να έχει αντίκτυπο ε, και στην αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης ε, της επικράτειας αλλά και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και να πω και κάτι γρήγορα για τα προγράμματα έρευνας όταν εργαζόμαστε με γεωργούς και έχουμε συμμετοχικές έρευνες, πρέπει να προσπαθούμε να ξέρουμε πριόρι που θέλουμε να φτάσουμε, γιατί μπορεί να αλλάξει η γνώμη ο γεωργός, πρέπει να είμαστε ε, ουσιαστικά ευέλικτοι, γιατί υπάρχουν περιορισμοί από τους γεωργούς και θα πρέπει να γράψουμε το σχέδιο της έρευνας, τα αποτελέσματα και στην πραγματικότητα θα πρέπει στην επιλογή των φακελών να επιλέγουμε τη μέθοδο παρά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα με γεωργούς ακόμη και αν δεν ξέρουν που πάνε. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε καινοτομίες που τελικά είναι πιο χρήσιμες για τους γεωργούς. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μορέλ, καθώς επίσης και τους άλλους δύο παρεμβάντες. Ε, μπορεί να αρχίσει τώρα η συζήτηση. Δύο λεπτά βέβαια αναπαρέμβαση και με την παράκληση να σέβεστε τον χρόνο που σας παρέχω. Η κυρια Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ πρώτα-πρώτα για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και οι τρεις μου, μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή στην χρήση ενέργειας μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία των Γιώργων και ποτέ με αντίθεσή τους. Θα σας ερωτήσω και ιδίω σχετικά με το παράδειγμα της Ουγγαρίας. Μιλούμε για την ανάγκη χρήσης της ηλιακής ενέργειας, της ε, αιωλικής ενέργειας, βεβαίως του βιολογικού καυσίμου. Τα είπατε και σε αυτά πράγματα. Αυτές τις ενέργειες πρέπει να μπορούμε και να τις αποδικεύουμε. Υπάρχουν όντως τεχνικές που μπορούν να αποθηκεύσουν το μεθάνιο που παράγεται από την ε, κατάσταση παραγωγής βιολογικού αερίου και το οποίο δεν είναι καθαρό ακόμη. Μπορεί να καθαριστεί λοιπόν σε εγκαταστάσεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι γεωργοί να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή. τον τομέα των καυσίμων πρώτης γενεάς για μένα είναι σημαντικό να παράγεται όχι μόνο η ελαιοκράμβη και το έλαιο που παράγεται από αυτήν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικούς ελκυστήρες, αλλά και πολλά λευκοματούχα τρόφιμα, τα οποία είναι σημαντικά για την διατροφή των αγελάδων μας, ώστε να εξαρτώμεθα λιγότερο από τις εισαγωγές. Άρα, αποτελεσματική χρήση των πόρων και προστασία απέναντι στην αλλαγή του κλίματος θα γίνει με τη συνεργασία της Γεωργίας μόνο εφόσον υπάρξει διαβούλευση με την ε, Γεωργία, εκπαίδευση των Γεωργών. Και έχω και την ερώτηση προς, ε, μια ερώτηση για τις ε, γαλλόφωνες παρεμβάσεις. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα μοιραστεί εδαφός στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Νομίζω ότι μπορούμε στον τομέα της κοινής αγροτικής πολιτικής να επιτύχουμε ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων ώστε να ενισχυθούν αυτές δηλαδή και οι μικρομεσαίες γενικότερα. Ευχαριστώ κύριο ε, Ρούπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τους καλεσμένους μας που πραγματεύτηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα και μας έδωσαν και ωραία παραδείγματα. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά για το μέλλον μας και θα πρέπει να τα λάβουμε δεόντως υπόψη κατά την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σίγουρα θα πρέπει να ζητήσουμε και τη γνώμη των γεωργών και να εξετάσουμε από κοινού μαζί τους κάποια πιλωτικά προγράμματα. Διάβασα πρόσφατα μία μελέτη Αμερικανών επιστημόνων με θέμα τη χρήση των λιμάτων και της ανακύκλωσης ε, των λιμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο. Ήταν ενδιαφέρον να έχουμε κάτι αντίστοιχο γιατί αν αποβεί αποδοτικό το ε, αμερικανικό μοντέλο, θα μπορούσαμε να το μιμηθούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα λίματα για να παράγουμε ε, καύσιμα. Όπως χρησιμοποιούμε απόβλητα τροφίμων, απορρίμματα τροφίμων ε, για να φτιάξουμε καύσιμα. Και σίγουρα η νέα γενιά καυσίμων θα είναι αυτή που θα παράγεται από τέτοιου είδους πρώτες ύλες. Ποια είναι η γνώμη σας, έχει κάποιο μέλλον ε, μια τέτοια πρόταση για να δημιουργήσουμε μια νέα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα ελλείμματα. Ευχαριστώ κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσει, γιατί πολύ συχνά ερχόμαστε εδώ και ακούγαμε για τι κρίσει των ΑΒ τομέα και το τι θα κάνουμε γι' αυτό. Και μερικέ φορέ ακούμε κάποια πολύ θετικά νέα. Ο κύριος Μορέλ, για παράδειγμα, μας έδωσε πολύ θετικές ειδήσει. Και η δήλωση που έκανε ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις παίρνουν περισσότερα κονδύλια από τις μικρές και περισσότερες επιδοτήσεις. Αυτό προέκυψε από όλες τις παρεμβάσεις και αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο, στη, τους αγρότες στη γη τους και αν έχετε θετικά παραδείγματα θα πρέπει να τα μιμηθούμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του κ. Γκλάτφελντερ για το βιοαέριο και την αναεροβική πέψη, Ποιε είναι οι ε, πιθανέ αλλαγέ που προτείνεται στον κανονισμό για τα λοιπάσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κλείσουμε καλά τον κύκλο. Γιατί είναι τεράστια αυτή η πρόκληση, κυρίως για τους Ελλαδούς ε, γεωργούς. Ε, και κτηνοτρόφου για την ε, παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπάρχει πίεση για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Και έχουμε παραδείγματα σχεδίων με αναεραβικούς, ε, αναεραβικούς μηχανισμούς μικρής κλίμακος που φαίνεται ότι έχουν δουλέψει στις κάτω χώρες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις ε, πιέσεις που υφίστανται οι γεωργοί. Κύριε Γκλάτφελντερ, λοιπόν, εσείς τι γνώμη έχετε για τις προτινόμενες ε, τροποποίησεις στον κανονισμό για τα λοιπάσματα. Πάντως, ε, πραγματικά, ακούγοντας τον κύριο Μορέλ και τον κύριο Μπαρέ, δημιουργήθηκε κάποιες θετικές σκέψεις και κάποια ελπίδα ότι μπορούν να οι γεωργοί να επιβιώσουν με την γεωργική δραστηριότητα. Γιατί μια πρόκληση είναι να ψητήσουμε τον κόσμο, να θρέψουμε τον κόσμο. Αν θέλω όμως σοβαρά να το κάνουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε να παραγάγουμε όπλα που σκοτώνουν τον κόσμο και τα κονδύλια αυτά της, ε, ε, που αφιερώνουμε στην αμυντική βιομηχανία να τα αφιερώσουμε στην παραγωγή τροφίμων γιατί αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό αγαθό από τα όπλα που σκοτώνουν κόσμο. Ο κύριος Άγνιο. Εδώ μιλάμε για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και τη γεωργία. Και ενώ αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυμητό για την εξοικονόμηση ενέργειας, ε, αυτό ε, τώρα αναφέρεται ότι θα βελτιώσει και τον κόσμο. Όμω δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν ε, θέλετε ε, ουσιαστικά να βελτιώσετε την κατάσταση, ουσιαστικά είναι η άντληξη διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει έλλειψη διοξιδίου του άνθρακα στην ε, ατμόσφαιρα για την ε, βέλτιστη καλλιέργεια του φυτού. αυτής. οι δεξαμενές χώνευση ή αναερόβιε είναι πολύ καλές. Αν μπορούμε ουσιαστικά να τις χρησιμοποιήσουμε όμως θα χρειαζόταν, παραδείγματο χάρη, να μετακινηθούμε κατά χιλιόμετρα και να πληρώνει ο καταναλωτής και αυτό είναι τρέλα. Εγώ προσπαθώ να βρω κάποιον ε, στον οποίο θα μπορούσα να πουλήσω το πάνελ μου ε, γιατί ε, δεν μπορώ να βρω κανένα που θα μπορούσε να το κάνει για μένα ενώ αν χρειαζόταν κάποια επιδότηση κάτι θα γινόταν. Επίσης πρέπει να διαφωνήσω με τον τρόπο που αναφέρεται για την πρόοδο. Τελικά νομίζω ότι οι φτωχοί θα πληρώσουν το κόστος. Επίσης αναφερθήκατε στην εξοικονόμηση ενέργειας ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να της αρέσει το γλυφοσάτ. Επίσης, ε, οι άνθρωποι θα, αν έπρεπε να πληρώνονται ουσιαστικά αξιοπρεπώς θα ήταν πολύ ακριβά τα τρόφιμα. Θέλω να ρωτήσω επίσης ε, για τις τάσεις σας ε, για τα απόβλητα ανθρώπων γιατί αυτά μπορεί να γίνουν λοιπάσματα για τις επόμενες σοδιές όμως πολλοί άνθρωποι φαίνεται να τα αποστρέφονται. Σας ευχαριστώ. Κύριος Έντρους. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Γεωργία που να ε, κάνει εξοικονόμηση πόρων ε, είναι σωστό ο στόχος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ωστόσο μεγάλες αποκλήσεις ανάμεσα στις 15 παλές χώρες της Ένωσης και τις νέες. Κύριε Κλάτφελντερ, πώς βλέπετε το δυναμικό της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και πώς, τι μάλλον τι πρέπει να γίνει ώστε να ενισχυθεί αυτό. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την συζήτηση και νομίζω ότι είναι πολύ αναγκαίο που γίνεται διότι η πτυχή της ενέργειας είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει πολύ τις τελικές τιμές των γεωργικών προϊόντων, διότι στο κάτω της γραφής όλοι είμαστε καταναλωτές πρώτα-πρώτα. Θα ήθελα να μιλήσω για τα συστήματα άρδευσης στην γεωργία, που μου φαίνεται πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζουμε ότι εφόσον αρδεύονται σωστά τα εδάφη, αυξάνεται η παραγωγή και ε, όλα πάνε καλύτερα. Ωστόσο υπάρχουν ε, προβλήματα σχετικά με την άρδευση στο, στα ευρωπαϊκά εδάφη και όλα αυτά έχουν σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεται, είτε ηλεκτρική είτε ενέργεια που προέρχεται από πετρέλαιο ή δίζελ. Και έχω λοιπόν την εξή ερώτηση. Έχετε λάβει υπόψη σας τον ενεργειακό παράγοντα ε, στον εξελεκτρισμό των συστημάτων άρδευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλικία ενέργεια για ε, την άρδευση. Ο κ. Άγνη μίλησε προηγουμένως για την έλλειψη ηλιακής ενέργειας σε ορισμένες περιόδους του χρόνου. Εγώ νομίζω ότι η ηλιακή ενέργεια δεν χρησιμοποιείται αρκετά στην ε, ε, γεωργία. Η ηλιακή ενέργεια δεν αρκεί βέβαια για να ε, κατεβάσει τις τιμές. Είναι όμως ένας πόρος πολύ προσιτός που δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. η ηλιακή ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα και την άρδευση αλλά και τις διαδικασίες αποξήρανσης. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες χρήσεις της ηλιακής ενέργειας στην Γεωργία. Αυτό θέλω να μάθω. Ευχαριστώ. Μαγκίνες, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για τις συνεισφορές σας. Για την πρώτη παρουσίαση Καλώ ήρθατε και πάλι. Πολύ καλά που σα βλέπουμε εδώ μεταξύ μα. Είπατε ότι μπορεί να είναι εμπόδια οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόεδρο. Μπορείτε ίσω να είστε πιο συγκεκριμένο για το πώ μπορούμε να του αλλάξουμε και πού. Και επίση, ε, τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη χωρί ευρωπαϊκή καθοδήγηση για να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Για να προχωρήσω τώρα Νομίζω ότι δεν βοηθάει η συζήτηση για ε, το να θέτουμε την ε, μικρή έναντι της μεγάλης γεωργίας, την, ε, την εκτατική έναντι της μικρότερης κλίμακας. Είναι πολιτική η συζήτηση αυτή και έχουμε πολύ μεγάλους γεωκτήμονες που θα μπορούσαν να δώσουν γη για την βιοπικιλότητα θα ήθελα να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την εξοικονόμηση των πόρων και την καινοτομία και αυτό είναι ακριβώς ο τίτλο της συζήτησή μας και ακόμη δεν ακούσαμε ποια είναι η έρευνα που γίνεται στον τομέα και αν έχουμε την ικανότητα στα κράτη-μέλη προκειμένου να πάει η γνώση στους γεωργού. εκεί όπου τη χρειάζεται γιατί οι γεωργοί ε, έχει νόημα να είναι αποδοτική ως προς τους πόρους και υπάρχει και ένα στοιχείο που νομίζω ότι είναι προβληματικό σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, πραγματικά ενθουσιάστηκα με την ιδέα των πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων ε, και επίσης έχουμε και την ε, ιδέα του care farming και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνία. Αυτές οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις ουσιαστικά είναι η απασχόληση γιατί ε, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχουν και άλλο εισόδημα και αν όχι, ποιος είναι ο μέσος όρος του εισοδήματός τους και ουσιαστικά τι θα επέτρεπε στους ανθρώπους αυτούς να ζουν από αυτή τη δραστηριότητα, να έχουν ένα εισόδημα δηλαδή. Σας ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Άουσλινγκ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ε, κύριε Κρατφέλτερ, είναι γνωστό ότι έχετε πολύ θετική άποψη για τα βιολογικά καύσιμα. Τώρα στη Γερμανία έχουμε συγκεντρώσει 15 χρόνων εμπειρία. Προ 15 χρόνων είχα, 15 ετών δηλαδή, είχα και εγώ πολύ θετική άποψη. Όμως τα τελευταία 15 χρόνια έδειξαν πως η χρήση του καλαμποκιού και μάλιστα σε ορισμένες περιοχέ καλλιεργούνται 50 και 60% των χωραφιών. Οικολογικά λοιπόν είναι μεγάλη ζημιά και ο οικολογικοί απολογισμοί τελικώ είναι ε, πολύ προβληματικοί. Ε, θα πούμε λοιπόν ότι όντω πρόκειται για μια γνήσια εναλλακτική επιλογή διότι ε, όταν καλλιεργώ καραμπόκι σε όχι απόλυτα κατάλληλα εδάφη έχω και πολύ ε, σημαντική εκπομπή διοξιδίων του άνθρακος. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και για την ελαιοκράμβη η οποία κράμβη χρησιμοποιείται ε, ε, στις ε, εναλλαγές σπορών μέχρι και 13% και αυτό χρειάζεται κάποια στιγμή να το σκεφτούμε τη χρήση για παράδειγμα ξύλου τη χρήση των αποβλήτων των βοηδών κοπράουν κλπ. να χρησιμοποιηθούν και αυτά, να προωθηθούν ως πηγή ενέργειας. Τώρα για την εξέλιξη στη Γεωργία. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας κύριε Μωρέν που είπατε ότι δεν πρέπει να κινηθούμε μονάχα σε προσυκολογική ε, και κατεύθυνση. Έχουμε πόρους όπως φωσφορούχα τα οποία κάποια στιγμή θα τελειώσουν και άλλοι πόροι ε, είναι πεπερασμένοι. Και το άζωτο επίσης που χρειάζεται ε, για να παραθεί πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργεια. Για ένα κιλό αζώτου χρειάζεται δύο λίτρα ε, καύσιμο. Άρα χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η χρήση των πόρων αυτών και να αντικατασταθούν από άλλους. Σας ευχαριστώ κύριε Χόισλινγκ. Κυρία Νόιχολ. Ganz herzlichen Dank. Ich habe keine Frage, aber ich habe zwei Gedanken, die äh, ich einfach unterstützen möchte. Herr haben... Δεν έχω ερώτηση. Έχω δύο σκέψεις που θέλω να θέσω υπόψη. Σας είπατε ότι ε, κάποια στιγμή θα πρέπει και η πολιτική ε, να σκεφτεί ορισμένα πράγματα. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να λυθούν αποφάσεις. Δηλαδή μας έχουν δώσει ένα ρόλο, αυτόν πρέπει να παίξουμε και πάνω εκεί μόνο βασιζόμαστε γιατί υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος. Σας ευχαριστώ πολύ διότι πρώτον καταστήσατε σαφές ότι η πολιτική αποφασίζει και μπορεί να αλλάξει και αποφάσεις, αλλά όχι μόνο και κάθε γεωργός μπορεί να αποφασίσει και μπορεί να επιλέξει διαφορετικές οδούς. Πρόκειται για απρόλυτα ε, ε, στοιχειώδη πράγματα που καμιά φορά τα λησμονούμε και κάνουμε σαν να μην υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Και η δεύτερη φράση που είπατε, είπατε καθαρά ότι δεν ζητούμε αύξηση παραγωγής απαραίτητα, όχι απαραίτητα μεγαλύτερες εσοδίες. Και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ορισμένοι θεωρούμε ότι πρέπει να ταΐσουμε τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε όλο και αποδοτικότεροι, όλο και παραγωγικότεροι, διότι εμείς εδώ η Ευρώπη δηλαδή πρέπει να ταΐσει ολόκληρο τον κόσμο. Όμως στο τέλος του λογαριασμού, τι θα κάνουμε με τη γεωργική μας πολιτική. Δεν είναι μοναχά η αύξηση της παραγωγής. Είναι όταν θα κάνουμε τον τελικό λογαριασμό εάν έχουμε ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Δηλαδή αν έχουμε φροντίσει και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό να επανερχόμεθα διαρκώς στην αντίληψη ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να προσπαθούμε να ταΐσουμε τον κόσμο ολόκληρο και να κρατήσουμε τα χέρια μας μακριά από τις γέες των άλλων, διότι οι ορισμένοι είναι γνωστό ότι προβαίνουν και σε αρπαγές γεών. Χρειάζεται λοιπόν ε, αυτοσυγκράτηση. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και τις ερωτήσεις σας που έδειξαν και πόσο ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις σας. Θα δώσω λοιπόν τρία λεπτά στον καθένα σας. Λοιπόν, πολύ είναι κάπως ε, σύντομος ο χρόνος, αλλά για να δώσετε κάποια στοιχεία απαντήσεων στις ερωτήσεις που σας υποβλήθηκαν. Δυστυχώ αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν εδώ στο Κοινοβούλιο και καμιά φορά οι συζητήσεις ε, χρονικώς περικόπτονται. Θα αρχίσω λοιπόν με σας κύριε Μπέλα Γκλατφέλτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ θερμός να μου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Θα προσπαθήσω πάντως ε, να χρησιμοποιήσω το δυνατόν καλύτερο τον χρόνο. Στα δέκα χρόνια που ήμουν μέλος στην Επιτροπή σας δεν μπόρεσα να μιλήσω δέκα λεπτά όπως μπόρεσα πριν. Τώρα θα προσπαθήσω να μιλήσω μόνο σε τρία λεπτά. Το θέμα του βιολογικού καυσίμου που σας απασχόλησε και στις ερωτήσεις σας. Εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο να παράγεται από ε, ανανεώσιμες πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το βιολογικό αέριο. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, συντάξει σχετική έκθεση η οποία έχει ταχθεί υπέρ της ιδέας αυτής. Για την χρήση του βιολογικού καυσίμου, του βιολογικού αερίου δηλαδή, το ερώτημα είναι τι γίνεται με την υπερβάλλουσα θερμότητα. Ε, το χειμώνα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ε, πλεονάζουσα αυτή θερμότητα για τη θέρμανση κατοικιών και καταστάσεων. Τι κάνει όμως το καλοκαίρι, θα χρειαστεί να ε, το σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αποθηκευτεί. Για, αυτά για το βιολογικό αέριο, για το βιολογικό καύσιμο. Υπάρχουν πολλά υποπροϊόντα, για παράδειγμα λεύκομα. Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, μου τέθηκε μια ερώτηση ένα ερευνητικό ε, ίδρυμα μελέτησε πόσα απόβλητα καταλήγουν στα νερά. Φτάνουν στο, στους σε πολλούς τόνους και ε, εάν υπολογίσει κανείς ότι ε, ο εγγουρικός πληθυσμός είναι το 2% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού και παρόλα αυτά ε, υπάρχει μια υψηλή αξία η οποία τελικώς καταλήγει στα απόβλητα νερά, σκέφτεται κανείς ότι θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια. Εγώ έχω ένα γνωστό ο οποίος χειρίζεται μια εγκατάσταση βιολογικού αερίου η οποία αποδίδει, αλλά τα υποπροϊόντα της εγκατάστασης βυθίου, δυστυχώς δεν έχω πλέον τις διαφανειές μου να μπορέσω να σας τις δείξω, τα υποπροϊόντα που είναι που είναι αυτή η, η λάσπη των αποβλήτων των βοηδών είναι σχεδόν υγρή. Δεν μπορεί όμως την εποχή αυτή του έτους να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα στα χωράφια. Άρα θα πρέπει κάπου να μπορεί να αποδικευτεί. Και τελικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάσταση τον χειμώνα διότι τα απόβλητά της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Το ίδιο με τις στάχτες που προκύπτουν από, τις, ε, από την χρήση των αποβλήτων για καύση. Οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούνται για ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος χαρακτηρίζουν τα αποβλητά τους, τη στάχτη τους δηλαδή, ως ε, βιολογικό απόβλητο. Οι μικρέ εγκαταστάσει όμως δεν μπορούν να το πράξουν αυτό και μπαίνουν σε δυσκολίε. Τώρα, εάν όντω μέσα στις τάχτε αυτές περιέχονται όλες αυτές οι θρεπτικέ ουσίες που μπορούν να διοχετευτούν πάλι στο έδαφος όπως άζωτο κλπ. Θείο. Πρέπει να ανακυπλώνεται και η στάχτη. Άλλη ερώτηση ήταν σχετική με την χρήση του διοξιδίου του άνθρακος σε θερμοκήπια. Θα ήταν όντως χρήσιμο να μπορούν να θερμαίνονται τα θερμοκήπια με τέτοιες ενέργειες και να μπορεί να διοχετεύεται και σε αυτά και ε, το διευθυντήτου του άνθρακος. Αλλά με τη γεωθερμική ενέργεια συχνά καταλήγει στην επιφάνεια και ε, διοξείδιο του άνθρακος ή άλλα αδρανή αέρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άρδευση. Εδώ το θέμα της ενέργειας παίζει υποδέστερο ρόλο. Κυρίως εδώ ρυθμίζει τα πράγματα η οδηγία ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Αυτό για μας στην Ουγγαρία είναι ένα πρόβλημα. Εάν δεν μπορούμε να αρδεύουμε για ορισμένες ημέρες διότι δεν μας επιτρέπει η οδηγία χρήση των υπόγειων νερών σε αυτά εγώ έχω κάνει και μια μελέτη να σας το πω αλλιώς που είναι το, το αποτέλεσμα της μελέτης λέει ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται τελικώς καύσιμο δίζελ για τις ε, αντλίες της άρδευσης παρά να μπαίνουν στα χωράφια συλλεκτήρες ηλιακής ενέργειας. Και τώρα μια παρατήρηση σχετική με τη Γερμανία. Τα λέω αυτά προς την κατεύθυνση του κυρίου Χόσλινγκ, όπου υπάρχουν 6.000 εγκαταστάσεις βιολογικού αερίου που χρησιμοποιούν και κοπριάγος, καύσιμο και άλλα. Η λύση θα ήταν λοιπόν μόνο το ποσοστό εκείνο ενέργειας να ενισχύεται με οικονομικά, με οικονομικά κίνητρα δηλαδή που χρησιμοποιούν ε, διάφορα είδη απόβλητων της κτηνοτροφίας. Αυτό θα ήταν καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει, ξεπεράσατε λίγο το χρόνο, αλλά το περιεχόμενο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λυπούμε που πρέπει να είμαι τόσο αυστηρό, αλλά έχουμε κάποιους κανόνες που οφείλουμε να τηρήσουμε. Κύριε Μπαρέ, ε, υπολογίζω στη δική σας ικανότητα σύνοψης ε, για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Καταρχήν, θα σας μιλήσω για την παρούσα κατάσταση. Ε, καταρχήν, η παρούσα κατάσταση υπακούει σε, ρόλους, σε ε, νόμους της φύσης και είναι τα πολιτικά συστήματα και πολιτικές αποφάσεις ε, που επηρεάζουν την λειτουργία της αγοράς. Γίνονται κάποιες επιλογές και γι' αυτό είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ο τρόπος που προσδιορίζουμε σήμερα την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σε μεγάλο βαθμό δεν προσδιορίζεται η αποτελεσματικότητα από τους γεωργούς, αλλά από τους ε, μεγάλες αλυσίδες ε, ε, διανομής και το διεθνές εμπόριο. Ε, τον τρόπο ρύθμισης τη χαλακτοκομικής αγοράς, ε, τη χρήση, την παραγωγή ελαιούχων σπόρων. Αυτοί καθορίζουν την αποδοτικότητα και όχι οι ίδιοι Και μάλιστα, δεδομένου των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων για την υγεία, που δεν, αναφέραμε καθόλου, θα πρέπει να με σωλικούς συμπέρασμα θα πρέπει να αλλάξουμε την προοπτική μας. Και όταν λέω να αλλάξουμε την προοπτική, πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα σενάρια. Καταρχήν έχουμε ένα σενάριο που λέει συνεχίζουμε την παρούσα πορεία και είναι το πιο εύκολο σενάριο γιατί ακολουθεί τη φυσική πορεία. Το θέμα είναι αυτό το σενάριο να μπορεί να μας επιτρέψει να, χρησιμο... να τηρήσουμε την ατζέντα του 21ου αιώνα σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων, την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, και την ε, τις παγκόσμιες επιστημιστικές ανάγκες. Δυστυχώς ε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ε, κατάλληλο αυτό το σενάριο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που προβλέπει κάποιες σημαντικές τομές και επίσης θα πρέπει να ανάλογα με το σενάριο που θα επιλέξουμε, να καθορίσουμε και την πολιτική και όχι να έχουμε βολοματικές πολιτικές που απλώς κάνουν κάποιες προσαρμογές. Και είναι σημαντικό και το θέμα της έρευνας, γιατί οι έρευνες κυρίως λαμβάνουν υπόψη τις ε, πολιτικές και γεωρικές καταστάσεις που είναι ισότιμες, ενώ θα πρέπει να γίνουν έρευνες και για εναλλακτικά σενάρια. Θα πρέπει να γίνει ελεγχός και εξακρίβωση και άλλων σενάριων, όχι μόνο του σημερινού. Θέλουμε σενάρια που θα είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα από κάθε πτυχή. Και Επίσης, για το χαμηλότερο εισόδημα που έχουμε σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ναι, θα πρέπει οι γεωργοί να έχουν δικαίωμα απόφασης, κάτι που δεν ισχύει, γιατί δεν έχουν ε, αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. Βρίσκονται σε ένα σύστημα που τους εμποδίζει να λάβουν ήδη τις αποφάσεις τους. Επίσης, το θέμα της άρδευσης. Εκεί έχουμε δύο διαφορετικές ε, προσεγγίσεις του μοντέλου. Καταρχήν βρέχει πρόθεσμη, ε, με σταθερές συνθήκες ε, και με αυτό, με αυτό το σενάριο μπορούμε να έχουμε αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον αντίκτυπο. Γιατί το παρόν σύστημα δεν δημιουργεί πολλές ε, προοπτικές, ενώ μέσω και μακροπρόθεσμα θα χρειαστούμε άλλα συστήματα, συστήματα σαν αυτά που μας παρουσίασε ο Κέβιν, συστήματα που προϋποθέτουν μεγαλή, πιο κυκλική οικονομία, καλύτερη κατανομή των εισοδημάτων καθ' όλη καθόλου το μήκος αλυσίδα αξιών και να δούμε τι χρειαζόμαστε και μακροπρόθεσμα. Που χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα έχει όχι μόνο ένα ε, μοντέλο ε, έντασης στη χρήση των πόρων, αλλά ε, μια μεγαλύτερη ε, φιδωλότητα στη χρήση των πόρων. Γιατί δεν θα έχουμε εσάι ε, άπειρου πόρου. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε το σύστημα, κάτι που είναι πιο δύσκολο και θα είναι και πιο χρονοβόρο. Και επίση δεν θα πρέπει να το επιβάλλουμε αμέσω στου γεωργού, γιατί είναι πολύ επιβαρυντικό. Αλλά στο όραμα που έχουμε για τη γεωργία θα πρέπει και αυτό το σενάριο να το εξερευνήσουμε. Μάλιστα, μερικοί γεωργοί είναι ήδη έτοιμοι να το κάνουν και στη βιολογική γεωργία υπάρχει αυτή η δυνατότητα αναζήτηση ε, και διερεύνηση διαφορετικών λύσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει και η συμβατική γεωργία. Επίση, ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και τι έρευνε ε, για τη βιολογική γεωργία. Μέχρι στιγμή το επίπεδο χρηματοδότηση τέτοια έρευνα είναι πολύ χαμηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση δεν είναι η πόλωση, αλλά η εκπαραλλήλου διερεύνηση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων για το μέλλον. Ευχαριστώ, ο κύριος Μουρέλ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις αντιδράσεις σας. Θα επικεντρωθώ σε τρία θέματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω μέσα σε τρία λεπτά. Μιλήσαμε πολύ για την αποδοτικότητα και για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βιοαέριο, παραδείγματος χάρη, για να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα. Αλλά όπως είπε ο συνάδελφος, όταν σκεφτόμαστε με όρους ενέργειας, πρέπει να βρούμε και άλλες πηγές και άλλους τρόπους αλλά το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πού μπορούμε να μειώσουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε και σε ό,τι αφορά τι πρακτικές σε επίπεδο εκμετάλλευση, ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε και πρακτικές ε, οι οποίες καταναλώνουν πολλή ενέργεια και εκπέμπουν πάρα πολλές εκπομπές. Παραδείγματο χάρη, ξέρουμε ότι η άρρωση του εδάφους ε, καταναλώνει τρομερή ενέργεια και επίσης ε, ξέρουμε ότι με την άρρωση αυξάνουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου, γιατί τα αέρια που είναι στη γη απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, ε, ως προς τις πρακτικές υπάρχουν πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Το ίδιο για να πούμε πως έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο σημερινό σύστημα. Έχουμε μεγάλη ε, εκμηχάνηση της γεωργίας, ε, έχουμε πάρα πολλές επιφάνειες που δεν συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες συνδεδεμένες καλλιέργειες, δηλαδή κάποια φυτά που θα δεσμεύσουν την ηλιακή ενέργεια και κάποια πιο χαμηλά φυτά στο έδαφο που θα ε, συλλέξουν άλλου είδους ενέργεια. Δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα σε πολλαπλά στρώματα. Για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τις οποίε αναφέρθηκα, το εισόδημα της εκμετάλλευσης είναι το μοναδική πηγή εισοδήματος ε, για τον Γεωργό. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν άλλο επάγγελμα πριν και επιλέγουν να καλλιεργήσουν αυτές τις εκμεταλλεύσει. Σήμερα στη Γαλλία έχουμε 30% γεωργικών εγκαταστάσεων όπου έχουμε άτομα που δεν προέρχονται από το γεωργικό περιβάλλον και δεν ε, βρίσκουν ε, το χάρη ανθρώπους ε, για να καλυφθούν κάποιες θέσει. Εδώ μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν συστήματα που έχουν νόημα και να αλλάξουν τον κόσμο και βάζουν το όνειρό στη Γεωργία γιατί διαφορετικά ε, θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο οι εκτάσεις και οι άνθρωποι αυτοί θα χάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να διατηρήσουμε και το νόημα και την ηθική. Και νομίζω μου μένει και λίγος χρόνος ακόμη, θα αποφεληθώ λοιπόν σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρώπη, ότι αν ε, θέλει να αλλάξει τον κόσμο, είδαμε με τη σκόνη γάλακτος που εξήγαμε στην Αφρική πριν από τις ποσοστώσεις, ε, όταν ε, βλέπουμε ότι δημιουργούμε ανεργία σε αφρικανικές χώρες, έχουμε μεγαλύτερη μετανάστευση. Έτσι λοιπόν, να αφήσουμε τις οικονομίες εκτός της Ευρώπης να τα καταφέρουν μόνες τους για να μπορούμε να περιορίσουμε και το πρόβλημα της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, τρεις ομιλητές για τις ε, παρουσιάσεις τους ε, και για τις οξυδερκείς απαντήσεις και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την συζήτηση. κατε και σε θέματα τεχνικών αλλά και πολιτικής, σε θέματα μοντέλων, τίθεται και το θέμα της καινοτομία, αλλά και του γιατί και για το πώς χρησιμοποιούμε τα διάφορα μέσα για να έχουμε καινοτομία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και ταχύτατοι στις απαντήσεις σας, αν και πιστεύω ότι όλο αυτό μας αναστάτωσε. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης και θα καλέσω εδώ στο βήμα τον καθηγητή Χαρπάς και τον ε, κύριο Πάτρικ Γόρπς για τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν. Merci. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, στο δεύτερο τμήμα της ακρόασής μας, ε, που θα μας παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές ε, στον κόσμο. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνε ε, με το πρώτο μισό τη ακρόαση. 10 λεπτά στον κάθε καλεσμένο για να μα παρουσιάσει τη θέση του και μετά απαντήσει με την ομίγυρη. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον καθηγητή Σέναν Χάρπας. Δέκα λεπτά παρακαλώ και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται από μια μικρή χώρα που έχει συμβάλει με μικρά πράγματα. Όριστε την τομάτα κεράσι και μεταξύ άλλων και την στάγδιν άρδευση, την άρδευση με σταγόνες. Η Γεωργία είναι από, τα βιβλικά χρόνια κιόλα ε, υπόθεσή μας. Η χώρα μου, το Ισραήλ, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι έρημος. Ε, όπως ξέρετε, η ανάγκη είναι η μητέρα της ε, ε επινόησης των ε, εφευρέσεων. Δεν έχουμε και πολύ νερό για να το διαθέσουμε στη Γεωργία, ούτε και εφορεσιές οι ε, δε συνθήκες στην έρημο είναι σκληρές. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ε, καλλιεργήσουμε την έρημο πήγαμε στην στάγδιν άρδευση που σημαίνει ότι δίνουμε στο φυτό ακριβώς το νερό που χρειάζεται και ακριβώς σε κάθε φυτό. Έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ νερό. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να πετύχουμε ε, ανάπτυξη των φυτών και χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα στάγδιν άρδευσης για να κάνουμε κάτι που λέμε στα αγγλικά fertigation, δηλαδή να προσφέρουμε στο φυτό όχι μόνο ε, το νερό που χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από το νερό και τα λοιπάσματα που χρειάζεται. Και μας επιτρέπει αυτό να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο νερό, διότι το νερό πηγαίνει κατευθείαν στις ρίζες του φυτού. Δεν ε, ε, διοχετεύεται στο υπόλοιπο του εδάφους. Γι' αυτό και είμαστε ηγέτης και σε αυτή την υπόθεση στο ανά τον κόσμο και μάλιστα ανακυκλώνουμε το 80% του νερού μας. Με αυτή τη στάγνη άρδευση και τη χρήση του συστήματος αυτού καταφέραμε να ανθίσει η έρημος. Και όπως βλέπετε στις ε, φωτογραφίες αυτές, βλέπετε μια ερημική περιοχή, μια περιοχή ερήμου δηλαδή, το 1959 και μετά όπου έχουμε 30 χιλιοστά ε, βροχή τον χρόνο, όχι την ημέρα ή την ε, ώρα. Και όπως βλέπετε εδώ στις άλλες φωτογραφίες μετά, καταφέραμε να ανθίσει η ερήμωση, διότι μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό με ε, πολύ λογικό τρόπο. Μάλιστα ακόμα και η δατοκαλλιέργεια κάνουμε στην έρημο, κάτι που θα σας φανεί εντελώς παράλογο, αλλά χρησιμοποιούμε το νερό από την υδατοκαλλιέργεια για να αρδεύσουμε τους, ε, τα φοινικόδεντρα που βλέπετε στο βάθος ε, της ε, φωτογραφίας κάνοντας έτσι μια βέλτιστη χρήση τα δε υποπροϊόντα της υδατοκαλλιέργειας, από τα ψάρια δηλαδή πάνε κατευθείαν στα ε, φοινικόδεντρα ως λίπασμα. Αυτό που λέμε καλλιέργεια ακριβίας είναι επίσης πολύ σημαντική. Χρησιμοποιούμε θερμική για να δούμε αν έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετό νερό ή αν το νερό ε, σπαταλάται. Χρησιμοποιούμε αυτές τις θερμικές κάμερες και μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς που βρίσκεται το πρόβλημα. Και έτσι πάλι μας επιτρέπει αυτό να εξοικονομούμε νερό και μας δίνει και τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε εάν η περιοχή μας που δεν είναι ομοιογενής αν αποδίδει τις ίδιες εσοδίε, διότι σε ορισμένες περιοχές, ορισμένα τμήματα δηλαδή της περιοχής, χρειάζεται περισσότερο νερό από άλλες. Χρησιμοποιώντας το σύστημα θερμικής απεικόνησης βλέπουμε ακριβώς που χρειάζεται περισσότερο νερό ή που ενδεχομένως χρειάζεται λιγότερο νερό από αυτό που δίνουμε, που προσφέρουμε στα φυτά. Χρειάζεται βεβαίως και να σκιάζουμε τα φυτά μας. Διαπιστώσαμε όμως ότι χρησιμοποιώντας δίχτυα διαφορετικής απόχρωσης έχουμε διαφορές στην ε, απόδοση. Βλέπετε ένα σύστημα εδώ που χρησιμοποιούμε δηλαδή διαφορετικών χρωμάτων σκίαστρα και δέστε τι γίνεται αν χρησιμοποιήσουμε στίχος μπλε ή ε, ε, κίτρινα δίχτυα στην περίπτωση του λούπινου. Βλέπετε τα λούπινα που ταυτόχρονα την ίδια, την ίδια ε, εποχή ε, δηλαδή φυτεύτηκαν και η κοπέλα που είναι δίπλα είναι η ίδια κοπέλα, δεν έχουν βάλει κάποια πιο ψηλή. Ε, η, η απόσταση, το ύψος των φυτών είναι πάρα πολύ μεγα, διαφορετικό, πολύ πιο, πολύ μεγαλύτερο και αυτό οφείλεται μόνο στη διαφορετική απόχρωση των δικτυών που χρησιμοποίησαμε και οι γεωργοί μας χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. Πώς διαπιστώνουμε, πώς να κάνουμε την βελτίωση των καλλιεργιών μας. Εμείς κατευθυνόμαστε στις ανάγκες των αγορών οι αγορές μας υπαγορεύουν τι θα πρέπει να διερευνήσουμε και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι καταναλωτές μας επίσης αλλάζουν όταν λέω οι καταναλωτές μας όταν λέμε οι πελάτες μας καλύτερα εγώ είμαι ερευνητικό κέντρο και πρώτα πρώτα οι πελάτες μας είναι οι γεωργοί στις δεκαετία του 1970 οι γεωργοί ήθελαν απόδοση σε ποσότητα μετά όμως μπήκαν στη, στο παιχνίδι και τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ ήθελαν τα φρούτα και τα λαχανικά να κρατούν όσο γίνεται περισσότερο στα ράφια τους. Κάναμε λοιπόν πολλές έρευνες για να αυξήσουμε τον χρόνο που αντέχει το φρούτο ή το κυπευτικό στα ε, ράφια. Χάσαμε βέβαια ε, στην πορεία αυτή κάποιο από το άρωμα και τη γεύση των φρούτων και των κυπευτικών. Έτσι, στη δεκαετία του 90 αυτό που μας ζήτησαν πλέον οι καταναλωτές είναι καλύτερη γεύση. Αλλά και καλύτερη εμφάνιση, εξωτερική εμφάνιση του φρούτου ή του κυπευτικού. Και τώρα οι ε, πελάτες μας είναι πλέον οι καταναλωτές και αυτό που θέλουν είναι διατροφική ποιότητα. Να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή διατροφική ποιότητα από τα προκυπευτικά που καταναλώνουν και ταυτόχρονα όχι μόνο να απολαύσουν το φρούτο ή το κυπευτικό αλλά να επωφεληθούν και από τα αντιοξυδοτικά, τις βιταμίνες που περιέχει το φρούτο ή και το λαχανικό. Ένα παράδειγμα μόνο, μίλησα πριν για τις ε, μικρούλες αυτές τομάτες που τις λέμε κεράσια. Έχουμε φτιάξει μια cherry tomato τώρα που έχει πολύ υψηλότερο επίπεδο καροτενοειδών και λικοπένης που προσφέρει αυτό το κόκκινο χρώμα στην ντομάτα η οποία λικοπένη είναι ένα θαυμάσιο αντιοξυδοτικό. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε την λικοπένη από την ντομάτα, την αφαιρέσουμε δηλαδή από την ντομάτα και να την προσθέσουμε σε άλλα είδη όπως είναι σοκολάτες, όπως είναι σόγια αυξάνοντας έτσι την αξία αυτών των άλλων ειδών διατροφής. Σε ό,τι αφορά την ζωική επιλογή, οι αγελάδες του Ισραήλ είναι αντικείμενο επιλογής εδώ και πολλά χρόνια. Πάλι το Ινστιτούτο μας αναμειγνύεται εκεί στην ε, γενετική προσπάθεια έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα σε μια κατάσταση όπου οι αγελάδες μας προσφέρουν 12.000 λίτρα γάλα τον χρόνο. Ε, το υψηλότερο, ε, η υψηλότερη ποσότητα σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο μέσω γενετικών μέσων, αλλά και με την επιλογή ποιοτική διατροφής για τις αγελάδες, ώστε να φτάσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο του γάλακτος, όχι μόνο ποσότητα αλλά και ποιότητα, σε ό,τι αφορά δηλαδή πρωτεΐνες και λίπη που ε, περιέχει το γάλα των αγελάδων. Ε, αυτών. Οι αγελάδες μας ε, μεγαλούν και σε ε, γεωργικές περιοχές, σε περιοχές ερήμου. Και έχουμε φτιάξει λοιπόν σταύρους οι οποίοι έχουν συστήματα με ανεμιστήρες και κατεωνισμό ύδατος πάνω στις αγελάδες, άρα είναι ένα είδος τζακούζι αυτό που τους κάνουμε μέσα στα υπόστεγά τους και αυτό πάλι τις βοηθεί να αποδίδουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος. Ακόμα δηλαδή και υπό συνθήκες ερήμου όπου οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλέ, αλλά μέσα στο, ε, στο οίκημα, μέσα στην εγκατάσταση, το σύστημά μας αυτό λειτουργεί σαν ε, ε, κλιματιστικό και διευκολύνει τις αγελάδες και τις κάνει να ζουν σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Η αγροβιοτεχνολογία μας επίσης ε, είναι σημαντική δουλειά για την αύξηση των ε, εσοδιών από τα περισσότερα φυτά. Η περισσότερη δουλειά που κάνουμε στρέφεται ή μάλλον γίνεται και στην βάση των περιορισμών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν έχουμε ε, ε ας πούμε εμπορικής εμπορικό επίπεδο παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποδόσεων. Ε, στα παλαιά χρόνια ένας γεωργός μπορούσε να, διατρέ... να διαθρέψει 15 ανθρώπους. Το 2007 είχε φτάσει στους 100 από έναν γεωργό. Το 2016 φέτος έχουμε φτάσει στον αριθμό των 200 ανθρώπων που μπορούν να τραφούν με τα προϊόντα ενός γεωργού. Και όλα αυτά βέβαια με την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργιών. Και αν εξετάσουμε τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν την ίδια τάση, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες οι άνθρωποι που διατρέφονται με τα προϊόντα ενός μονογεωργού είναι πολύ χαμηλότερος, από 2 έως 20 από έναν γεωργό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα είναι και η διατήρηση των γεωργικών μας προϊόντων μετά από την εσοδεία και με τεχνολογίες αποθήκευσης. Έχουμε φτάσει σήμερα σε μια κατάσταση όπου χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε 0,5% των σπόρων που χρησιμοποιούμε και αυτό γίνεται με επιστημονικά μέτρα τα οποία έχουμε λάβει και έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό απολειών στον κόσμο. Πολύ ευχαρίστως ε, διαθέτουμε τις πληροφορίες αυτές και σε άλλες χώρες και ιδίως βέβαια στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι μπόρεσα να σας ανοίξω λίγο τα μάτια στα όσα κάνουμε στη Γεωργία, στο Ισραήλ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε κύριε Άρπας. Πραγματικά πολύ εύστοχη οξυδερκής παρουσίαση και με αίσθηση του χιούμορ ταυτόχρονα. Περνάμε τώρα στον κύριο Πάτρικ Βόρμς για επίσης σε μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Θα ακολουθήσει, όπως είπα, συζήτηση με τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βάτησε και τον τίτλο του καθηγητού. Μακάρι να ήμουν, αλλά δυστυχώ δεν είμαι. Ήρθα να σας μιλήσω για την αγροδοσοκομεία που ε, δίνει μια όθηση στην παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα. Ε, δεν θα επισέλθω στη συζήτηση μεγάλων και μικροκαλλιεργητών ε, και ποιο ε, θρέφει περισσότερο το κόσμο. Το θέμα είναι τι εργαλεία χρησιμοποιούν. Έχουμε την έδρα μα στον Αϊρόμπι, κυρίω στι τροπικέ και υποτροπικέ ζώνε, αλλά και σε τη ζώνη. Γύρω στου 500 επιστήμονε έχουμε και εξετάζουμε το ρόλο των δέντρων στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Και το μέλλον θα πρέπει να παράγουμε πολύ περισσότερα τρόφιμα για να θρέψουμε τον πληθυσμό. Επίση, ε, πώ θα κάνουμε τι ιερικέ εκμεταλλεύσει ανθεκτικέ στι ακραίε καιρικέ συνθήκε ε, ενώ θα πρέπει να μειώσουμε ταυτόχρονα τι τεράστιε ε, εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου που παράγει και ο τομέα. Στο, στην άγρο δασοκομεία έχετε και το, τη δασοκομεία μέσα, οπότε θα η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή ενός δάσους. Βέβαια, έχουμε διαφορά μεταξύ ε, δάσους και δέντρων και δέντρων και ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Βλέπετε με συνδυασμό των δύο φωτογραφιών πόσο ένα χάρτη της παρουσίας δέντρων στον κόσμο και την κατανομή ανθρώπων στον κόσμο. Και ε, τα δέντρα δεν παρέχουν απλώς υλοτομικό υλικό ή καύσιμα, συμβάλλουν στην διατήρηση ανθρώπινης ζωής και στην γεωργία. Επίσης, ε, έχουμε εδώ τη συμπερίληψη αιωνόβιων φυτών και τις, εντάσσουμε τέτοια είδους ε, φυτά στην ε, γεωργική παραγωγή, στις γεωργικές Εδώ έχουμε μια δοσόδη περιοχή στη Γαλλία από τη δεκαετία του 50, ένα παράδειγμα στην Ισπανία, στις, στα λιβάδια με τα χείρο Πατανέγρα, και στο σύστημα αυτό, τα σύστηματα αυτά με παρουσία δέντρων είναι πολύ πιο αποδοτικά από τα συστήματα που χρησιμοποιούν τη μονοκαλλιέργεια. Επίσης, εδώ έχουμε το πιο αστείο παράδειγμα της αγροδασοκομείας, γιατί εδώ έχουμε Σρι Λάνκα, ε, ε παραγωγή Ινδικής καρύδας και επίσης ε, έχουμε και ψυχανθή που δεσμεύουν άζωτο στο έδαφος. Και επίσης ε, χρησιμοποιούνται τα απόβλητα στο τοπικό στάσιο παραγωγής βιομάζας. Τώρα, γιατί οι γεωργοί επιλέγουν την παρουσία δέντρων στα λιβάδια σας, στα χωράφια τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι εξυπηρετούν τα δέντρα με σημαντικές υπηρεσίες βιοσυστημικές. Βλέπετε εδώ ένα, μια περιοχή στη Ρωσία, στη Νότια Ρωσία, με εκατοντάδες χιλιάδες ε, του ίδιου τοπίου έχουμε ένα δίκτυο τέτοιων χωραφιών με πολλά δέντρα, συνήθως είναι λεύκες και άλλα και με η παρουσία των δεντρών ε, ακριβώς μειώνει την αποξήραση που προκαλούν συνήθως ισχυροί άνεμοι στην περιοχή αυτή. Επίσης, ε, τα δέντρα, οι ρίζες των δέντρων ε, είναι πιο βαθιές όταν από τις ρίζες των, των φυτών της καλλιέργειας. Οπότε ε, συμβάλλουν στην καλύτερη ε, δέσμευση του οργανικού άνθρακα στο έδαφος και χρησιμοποιούν ως και στις, χρησιμεύουν ως στις καλλιέργειες. Εδώ έχουμε μία στην αριστερή πλευρά ένα διάγραμμα που δείχνει ε, την απώλεια ηλιακού φωτός σε ένα ξερό, σε ένα χωράφι χωρίς δέντρα και στην άλλη περίπτωση έχουμε παρουσία των δέντρων στην ίδια, στο ίδιο χωράφι, με πολύ μικρότερη απώλεια του ηλιακού φωτός. Και όσο περνάει ο χρόνος θα διαπιστώσετε ότι η αύξηση, ε, ε, η αύξηση της αποδοτικότητας του, του ΣΥΤΟΥ μειώνεται στο μέτρο που ε, έχουμε λιγότερα φυλώματα, πιο ωραία φυλώματα στα δέντρα. Οπότε διαπιστώνουμε ότι ο Γεωργός δεν μπορεί να ε, περιμένει ίδια απόδοση σιτηρού όλα τα χρόνια. Θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ως δασοκόμος, γιατί ε, σίγουρα μερικές φορές ε, θα μειώνεται η παραγωγή του, αλλά η, η δασοκομική, το δασοκομικό τμήμα της παραγωγής αυξάνεται. Επίσης γνωρίζουμε τα προβλήματα που διάβρωσης εδάφους προκαλούνται από τις καταιγίδε. Αυτή τη διαδικασία την αναστέλουν τα δέντρα που συλλέγουν το νερό, εμποδίζουν τη διάβρωση και ε, δεσμεύουν το νερό στο υπέδαφος, ώστε να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ξηρασίας. Επίσης, εδώ έχουμε μετρήσει τον αριθμό των ρίζων που έχουν τα δέντρα σε ένα σύστημα δοσοκομείας και ένα σύστημα αγροδοσοκομείας. Και μάλιστα στο σύστημα δοσοκομείας ε, ε, οι, οι είναι σχετικά επιφανειακές, ενώ στο σύστημα αγροδοσοκομείας οι ρίζες είναι πολύ βαθύτερες. Και όταν έρχεται η ξηρασία στο σύστημα δοσοκομείας τα δέντρα υποφέρουν, ενώ στο σύστημα αγροδοσοκομείας τα ε, δέντρα συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Γι' αυτό και τέτοιου συστήματα που βλέπουμε πώς αλλάζουν μετά από 35 χρόνια, βλέπουμε ότι ε, παράγουν ε, πολύ χρήσιμο, ξύλο και βιομάζα, πολύ περισσότερο από ότι μόνο τα σοκομικά συστήματα. Επίσης, ε, πολύ, πολύ χρήσιμες οικοσυστημικές μελέτες δείχνουν ότι τα αγροδοσοκομικά συστήματα έχουν διπλάσια δέσμευση άνθρακα στο έδαφος. Επίσης, ε, είπαμε να ασχοληθούμε με παγκόσμια, μη ευρωπαϊκά παραδείγματα. Ένα σημαντικό ε, δείχνει ένα τοπίο τη δεκαετία του 80 στον Νίγηρα. Ε, παντελώς ε, ερημικό, τίποτα δεν φυτρώνει εκεί και μάλιστα μία περίοδο βροχών τεσσάρων εβδομάδων και όλος ο υπόλοιπος χρόνος είναι ζεστός και χωρίς νερό. Και εδώ χρόνια μετά, με μερικά χρόνια μετά έχουμε 5 εκατομμύρια ε, εκτάρια νέου ε, αγροδοσοκομικού συστήματος με 500.000 τόνους περισσότερο από πριν. Και μάλιστα τα δέντρα δεσμεύουν το άζωτο στο έδαφος και ξαναδίνουν το άζωτο αυτό λίπασμα στις καλλιέργειες. Και μάλιστα δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των νέων καλλιεργιών και των δέντρων και μάλιστα έχει δείξει έρευνα ότι σε αυτά τα 500.000 500 τόνους έχουμε αυτά τα 5 εκατομμύρια εκτάρια έχουμε 500.000 τόνους περισσότερο ε, τρόφιμα προϊόντα από πριν. Και μάλιστα στις περιόδους ξηρασίας ε, εξακολουθούν τα γεωρικά πλεονάσματα που χρησιμοποιούνται σε ε, άλλες περιοχές που δεν έχουν ακόμη μυθεί στην αγροδασοκομεία. Τώρα, αν λάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα ωφέλη της αγροδοσοκομείας και τα συνοψίσουμε, έχουμε το Land Equivalency Ratio και βλέπουμε ότι ε, ποια είναι η παραγωγικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα σύστημα αγροδοσοκομείας που, χρησιμοποιούν, που χρησιμοποιεί βιομάζα ε, για καύσιμο και είναι παραγωγή σιδηρών, βλέπουμε ότι ο λόγος ε, ε, ισοδυναμίας προς τη γη είναι ακόμα 43 που είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι δεν έχουμε απλό σύστημα γεωργίας ή απλό σύστημα δασοκομείας. Επίσης, εδώ βλέπουμε μία φάρμα στο Αγρομίσθωσης. αγρομίστοσης. Ε, φυσικά δεν μπορούσε σε τόσο σύντομη περίοδο της αγρομίστοσης να ασχοληθεί με τη δασοκομεία και υλοτομία και διάλεξε τα μήλα, τις μιλιές. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η καλλιέργεια και τελικά έχει 1,1 ε, ισοδυναμία γης ε, λόγω και 10% ε, αύξηση της παραγωγικότητας. Και αυτός ο λόγος όταν έχει καταμετρηθεί σε χώρες όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ 1,2 και 1,4. Βέβαια, σε, στον Νίγηρα είναι πολύ υψηλότερος αυτός ο λόγος. Τώρα, γιατί δεν καλύπτεται, αν είναι τόσο καλό, στην αγροδασοκομεία. Καταρχήν, είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα το αγροδασοκομικό. Και ένα συμβατικός γεωργό θα, αν δεν κάνει λάθο, χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία, του ίδιου πόρου και τον ίδιο εξοπλισμό, θα έχει ε, περίπου την ίδια απόδοση με του γείτονε. Ενώ ο αγροδασοκόμος, ο Γεωργό, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σαν δασοκόμος, που να ε, τα δέντρα, πόσο μακριά πρέπει να είναι, πότε να τα κλαδεύω και μερικές φορές ε, θα πρέπει να, κάνει, να πάει ακόμη πιο μακριά. Θα πρέπει να κλαδεύει όχι μόνο το φύλλωμα, αλλά και τις ρίζες για να μείνει έδαφος και για τις καλλιέργειες. Και έτσι οι γεωργοί που χρησιμοποιούν την αγροδοσοκομεία τελικά αυξάνεται, βλέπουν την αποδοτικότητά τους να αυξάνεται, αλλά οι περισσότεροι κάνουν λάθος, εκτός και να έχουν τις σωστές συμβουλές και έτσι η αποδοτικότητά τους θα μειωθεί. Είναι πολύ περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση και ακριβώς γι' αυτό ευνοεί τον μικροκαλλιεργητή και δείχνει ε, τον πίνακα αυτό της ΦΑΟ που λέει άσχετα από την καλλιέργεια και άσχετα από τη χώρα οι μικροκαλλιεργητές ε, είναι οι πιο αποδοτικοί. Όσο μεγαλύτερη είναι η γεωρική εκμετάλλευση τόσο λιγότερο αποδοτική είναι. Για τον απλούστατο το λόγο ότι οι μικροκαλλιεργητές ήδη ασχολούνται με τη γεωργία ακριβίας και χρησιμοποιούν τα καλύτερα εργαλεία γεωργίας ακριβίας που είναι το ανθρώπινο μάτι. Και τέτοιου είδου μικρέ καλλιέργειε παράγουν μεγάλα επίπεδα βιομάζα, έχουν μεγάλη αποδοτικότητα και επίση κρατούν την πυκνότητα του πληθυσμού για πολλού αιώνε. Αντίθετα, βλέποντα ένα χωράφι σαν αυτό, δεν βλέπω πρόοδο τη γεωργία, βλέπω μόνο ζημιέ και ε, απώλειε. Δεν χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα αγροδοσοκαμία. Ένα εδώ ε, δέντρα που κάνουν τη φωτοσύνθεση και χρησιμοποιούν το νερό που μπορούν μέχρι την περίοδο των βροχών να το χρησιμοποιήσουν. Επίσης, ο Γεωργός αυτός έχει καλή παραγωγή αραβοσίτου στο Μαλάουι, αλλά θα πρέπει να εργαστεί σκληρά, γιατί θα πρέπει ε, να προσέχει και τα δέντρα του, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί αν δούμε τις μετρήσεις, της αποδόσεις χωραφιών, έχουμε 36 χωρίς λιπάσματα, 213 χωράφια με λιπάσματα και ούτω καθεξής, βλέπουμε ότι η πραγματική αύξηση της αποδοτικότητας δεν οφείλεται, από τη χορή, δεν οφείλεται στη χορήγηση λιπασμάτων, αλλά στην προσθήκη δέντρων. Και μάλιστα αν βάζουμε λιπάσματα σε χωράφια που έχουν ήδη δέντρα, η διαφορά είναι ελάχιστη. Δεν λέω ότι είναι άχρηστα τα λοιπάσματα. Αλλά εδώ μιλάμε για απεμπλουτισμένα εδάφη που αυτό που ενδιαφέρει ε, για να είναι πιο γόνιμα είναι να έχουν μεγαλύτερη δέσμευση οργανικού άνθρακα και όχι περισσότερα τεχνητά λοιπάσματα. Τώρα, φινικέλο στη Βραζιλία. Μετά από μια πενταετία έχουμε αποδοτικότητα μεταξύ 6 και 9 τόνους ε, ανεκτάριο το χρόνο σε σχέση με τα, τους 5 τόνους ε, του γείτονα που έχει μονοκαλλιέργεια. Επίσης έχουμε πολύ περισσότερα φρούτα Έχουμε και προστατευτικέ καλλιέργειε, αντιδιαβρωτικέ μεταξύ των δέντρων και όταν οριμάσουν τα δέντρα θα έχουμε και υλοτομία. Οπότε πολύ πιο περίπλοκη ε, διαχείριση αλλά και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Και μάλιστα είναι σχεδόν διπλάσια αποδοτικότητα από την αποδοτικότητα της μονοκαλλιέργειας. Μια και ο χρόνο πιέζει να περάσω το τελευταίο επιχείρημα τη κλιματική αλλαγή. Είναι αδύνατο να αργεί στι νέε συνθήκε χωρί να συμβάλλει στο μετριασμό των κλιματικών συνθήκων και έχει ρόλο να διαδραματίσει. όπω και αν γίνει η καταμέτρηση, ε, η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 1 τρίτο των παγκόσμιων αερίων θερμοκηπίων στον κόσμο. Ε, ακόμη και λάβουμε υπόψη τη δέσμευση του άνθρακα. Και μάλιστα αυτό που δεν είναι προφανές είναι πόσα δέντρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όταν ε, έχουμε αποψήλωση. Τι αναδάσου θα πρέπει να γίνει. Στη φάση της ανάπτυξης των αγροδοσοκομικών συστημάτων έχουμε 1,5 γιγατόνους μετριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 1 τρίτο του συνολικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτή η λύση δεν είναι μόνιμη, γιατί από τη στιγμή που θορυμάζουν τα δέντρα δεν δεσμεύουν τόσο πολύ άνθρακα, αλλά και αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Τώρα, πώς ενθαρρύνουμε τους γεωργούς. Σήμερα οι γεωργοί χρησιμοποιούν περισσότερη την αγροδοσοκομεία, αλλά το, η διαχείριση είναι πολύ περίπλοκη. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να αναπτύξετε ένα σύστημα που δεν θα προσδιορίζει με ακρίβεια πόσα δέντρα χρειάζονται ένα εκτάριο και τι θα πρέπει να κάνει κάθε μέρα ο γεωργός, αλλά θα πρέπει να δώσετε κίνητρα στους γεωργούς να κάνουν το σωστό, πιο μακροπρόθεσμα. Και θα πρέπει να έχουμε ένα ε, τρόπο καταμέτρησης ε, του οργανικού άνθρακα στο έδαφος. Και με βάση αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καταμετρούμε την, τις προσπάθειές του και να δίνουμε τα κίνητρα. Αυτά και ελπίζω να συναρπαστήκατε όπως και εμείς από το δυναμικό αυτής της τεχνολογίας. Merci, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε και πάλι για τις ε, πολύ ωραίες παρεμβάσεις. Θα δω, ανοίξω τώρα τη συζήτηση και θα δώσω το λόγο στους να ρωτήσω και την Κομισιόν αν θέλει το λόγο. Κύριος ε, Λόγκο, στα πέντε λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας ε, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θεωρούμε ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων στην ε, οικονομία μας ε, ταυτόχρονα επιδιώκει και πολλαπλούς στόχους, ε, από τη μία την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του αντίκτυπου του περιβάλλοντος, χωρίς ε, να έχουμε μείωση της παραγωγής και επίσης να έχουμε και δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη. Η υποδοτικότητα των πόρων είναι μία από τις προτεραιότητες της Κομισιόν καθώς είναι ζωτική για την υλοποίηση των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Η αρχή βρίσκεται στην καρδιά μιας βιώσιμης γεωργίας και μιας αγροδοσοκομείας όπως εγγράφεται ήδη στην ΚΑΠ και έχει εγγραφεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου και βρίσκεται μεταξύ των πρετήτων. Η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι μια πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα και να επιτρέπει να στηρίξουμε όλα τα βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Γι' αυτό και είναι η γεωργική πολιτική δίνει τη δυνατότητα οι γεωργοί να επιλέξουν μοντέλα τα οποία κατά την άποψή τους θα είναι τα πιο σωστά. Η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες αναφέρθηκε και η καινοτομία είναι σημαντική προκειμένου να έχουμε αποδοτικότητα των πόρων ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο εκμετάλλευσης ε, ή στο σύνολο της γεωπιστικής αλυσίδας και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που τίθεται στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή γεωργία. Μόνο η γνώση μπορεί να μας επιτρέπει να έχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον το σύστημα της γνώσης στο γεωργικό επίπεδο θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό η έρευνα και η καινοτομία είναι σίγουρα προτεραιότητες. Με την διτή ευθύνη για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη αφενός και την γεωργική έρευνα και την καινοτομία αφετέρου, βλέπω με σαφήνεια τα πλεονεκτήματα και το δυναμικό συνεργειών, να σας να συνδέσουμε τις πολιτικές με τα μέσα, να συνδέσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και τον ορίζοντα 2020 το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εντάξουμε τα πολιτικά μέσα χρησιμοποιώντας ε, την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομίας αυτό φαίνεται να προωθεί σημαντικά την γεωργική καινοτομία και τον αντίκτυπο επιτόπου. Το να δημιουργήσουμε συνδέσμους, συνέργειε, συνεργασίες προκειμένου να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των πόρων στο σύνολο του επιστηστικού συστήματο είναι προτεραιότητα και νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Εμείς δεσμευόμαστε σε αυτό και ο κύριος Μπαρέ, ο καθηγητής Μπαρέ θα έχει την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να συμμετάσχει σε ένα workshop το οποίο οργανώνουμε. Και για να σεβαστώ και το χρόνο θα σταματήσω εδώ. Όμως θα ήθελα να σας ε, ανέφερα αυτά τα πράγματα για να σας πω ποια είναι η δική μας ε, πρόσληψη των όσων υπόθηκαν σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε ε, τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Έχουμε μόνο 10 λεπτά. Καταρχήν ο κύριος Μπέλτερ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το πάνελ για αυτές τις ενδιαφέρουσες και ενθουσιώδεις παρουσιάσεις. Έχω μία ερώτηση στον καθηγητή Χαρπάς. Αναφερθήκατε σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και από τη σκοπιά της επιστημονικής συνεργασίας. Τι θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε κάτι παραπάνω από τις βέλτιστες πρακτικές. Τι μπορεί να γίνει. Παραδείγματο χάρη για να καταπολεμήσουμε τις ζωνόσους. Και κάτι ακόμα, η καινοτομία έχει προχωρήσει πολύ πράγματι, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη. Τι σκέφτεστε γι' αυτό. Οι νέοι στη Γεωργία είναι ένα άλλο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της τεχνολογίας ενδιαφέρονται οι νέοι ιδιαίτερα για τις καινοτομίε κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα της γεωργίας. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγκτου. Ευχαριστώ. Ιδιαίτερα συναρπαστικέ οι παρουσιάσεις. Κάποιες ερωτήσεις, καταρχήν στον κύριο από το Ισραήλ. Με μόνο 30 ε, χιλιοστά ε, ουσιαστικά άρδευση στο χρόνο του στήθηκα από πού προέρχεται το επιπλέον νερό. Ξέρω ότι το, όταν το έχετε το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά έχετε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή στι αγελάδε και στον Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε ότι αν συνεχίσετε την οδό τη γαλακτοπαραγωγή, οι αγελάδε ε, μπορεί να παρουσιάσουν διάφορα προβλήματα, ε, δεν έχουμε μεγάλη αξία στο σφάγιο. Έχετε εσεί αυτά τα προβλήματα ή απλώ τα γνωρείτε. Και με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που είπατε ε, για τα γονίδια. Θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτή την επιτροπή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν αυτό το ε, ε, editing των γονιδίων ότι είναι επιβλαβές όπως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και θέλουν να το σταματήσουν. Στην Αφρική τώρα χρησιμοποιείται το χαρουπόδεντρο ε, μεταξύ ουσιαστικά στην αγροδοσοκομεία, μεταξύ των καλλιεργιών. Επίσης δεν θα μπορούσαμε όλοι να ακολουθήσουμε ε, την οδό του να φυτέψουμε μιλιές. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και σκέφτομαι ε, εδώ ουσιαστικά πώς ε, ουσιαστικά θα συλλέξετε τους καρπούς από τα δέντρα και ξέρω ότι είχα ε, στην Αφρική, ε, μεγάλη αγροδοσοκομεία, όμως ε, η μία δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν το πώς θα τεθεί σε εφαρμογή και θα συνεχιστεί. Και Επίσης, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή τη σύνθεση μεταξύ των δέντρων και της, των καλλιεργητικών εδαφών. Ευχαριστώ κύριε Άγνιου, κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δημιουργητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλές από αυτές τις ιδέες. Το Ισραήλ έχει πάει πολύ μακριά στο θέμα της έρευνας και της ε, τεχνολογίας και θέλω να ρωτήσω πόσα δαπανίσατε ε, προκειμένου να διαθέσετε αυτή τη γνώση στους αγρότες και να μπορεί να εφαρμοστεί. Και μία ακόμη ερώτηση έχει να κάνει με τα δέντρα και τη χρήση των ε, δέντρων ως μέσον παγίδευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Αν ε, δούμε τα κριτήρια ε, στο πλαίσιο της λούλους, της χρήσης γης, της αλλαγής της χρήσης της μπορείτε να δείτε αυτά τα κριτήρια ως ευκαιρία για την αγροδοσοκομεία ή θεωρείτε ότι το λούλους και οι σχετικοί παράγοντες είναι αρνητικοί και έχουμε και φυσικά και μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά ε, τους ελέγχους για την πολλαπλή συμμόρφωση. Αν ε, θα πρέπει να είναι ε, κάθε δέντρο μέρος των υπολογισμών, τότε έχετε δίκιο. Θα πρέπει να κάνουμε τα μαθήματά μας. Όμως, εσείς μιλήσατε και για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας που έχουμε αυτή τη στιγμή να προωθήσουμε τη συνεργασία στον τομέα αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερες ανησυχίες ε, ανησυχούμε ότι θα το καταπνίξει η γραφειοκρατία. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε κάποιες συμβουλές από τους εμπειρογνώμονες για να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία εκεί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους δύο καλεσμένους για τις παρουσιάσεις τους. Έχω μία ερώτηση για τον καθηγητή από το Ισραήλ, τον κύριο Χαρπάζ. Ε, σε ό,τι αφορά τη γαλακτοπαραγωγή. Έχετε μεγάλη γαλακτοπαραγωγή στο Ισραήλ και γνωρίζουμε ότι ε, το Ισραήλ ε, βρίσκεται στην αιχμή της ζωοτεχνικής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούμε πολύ για το θέμα αυτό της ε, πρωτεϊνικής διατροφής των ε, αγελάδων. Μερικοί είναι υπέρμαχοι της γενετικώς τροποποιημένης όγιας λόγω των πρωτεϊνών, άλλοι δεν θέλουν να χρησιμοποιούμε ε, τέτοιου είδους γενετικώς τροποποιημένης όγιας στην Ευρώπη. Βέβαια δεν την παράγουμε, οπότε αναγκαστικά την εισάγουμε. Εισάγουμε από την Αργεντινή για παράδειγμα, γιατί είναι αδύνατον να έχουμε παραγωγή γάλακτος χωρίς πρωτεϊνούχες ζωοτροφές στη διατροφή των αγελάδων. Εσείς πώς χειριστήκατε το θέμα. Μας μιλήσατε για την ανάπτυξη του κλάδου και μας είπατε ότι κάποια στιγμή τα σούπερ μάρκετ σας ζήτησαν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και σίγουρα η διάρκεια ζωής των τροφίμων είναι σημαντική για να αντέχουν περισσότερο στα ράφια, περισσότερο χρόνο στα ράφια, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της υγείας του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει μοναδικός μας στόχος να είναι το κέρδος των σούπερ μάρκετ. Εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε καταναλωτές, δεν είμαστε όλοι Γεώργοι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας χαρώ και να πω τον κύριο Χάρπας ότι χάρηκα που μου είπατε ότι κάνετε τζακούζι στις Αγελάδες και ότι ανακυκλώνετε το 80% των αλλημάτων. Επίσης έχετε ελάχιστη απώλεια των σιτηρών χάρη στον καλό τρόπο αποθήκευσης. Οπότε φαντάζομαι για να αναπτύξετε όλες αυτές τις τεχνολογίες χρειαστήκατε και πολύ χρόνο και πολύ χρήμα για να καταλήξετε σε αυτή την ισορροπημένη ανάπτυξη και στην ελαχιστοποίηση των απολειών. Ερωτώ λοιπόν, η πανεπιστημιακή κοινότητα πώς συνεργάστηκε με το γεωργικό κλάδο στο Ισραήλ και πόσο κόστισαν όλες αυτές οι επενδύσεις, πόσο, τι ποσοστό του προπολογισμού σας αφιερώνεται σε τέτοιου είδους επενδύσεις και σε τέτοιου είδους έρευνες. Επίσης, τεχνολογίες που αναφέρατε, τη στάγδινα άρδευσης, κατευθείαν στις ρίζες ε, ή η τεχνολογία αποθήκευσης ε, των ε, σιτηρών. Εφαρμόζονται όλες αυτές τις τεχνικές, αν το γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κάνετε εξαγωγή αυτών των τεχνολογιών ή βλέπετε δυνατότητα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μεταφέρετε την πλούσια αυτή τεχνογνωσία σας και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάρπας. Είχατε μια ενδιαφέρουσα διαφάνεια για το πώς ε, η παραγωγή των τροφίμων ε, κινούταν βάση των ετοιμάτων των καταναλωτών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν οι καταναλωτές απομακρύνθηκαν ποτέ από την γεύση και ε, αν είχε καλή γεύση ή όχι το φαγητό. Αν ο καταναλωτής ε, μας καθοδηγήσει για το μέλλον. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να δούμε στο μέλλον ε, το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων και δεδομένων το μεγέθους, του αριθμού των τροφίμων ε, που εξάγονται και η Ιρλανδία εξάγει αρκετά τι θα κάνετε αν ε, πει ο καταναλωτής έρχεται από πολύ μακριά το προϊόν αυτό, τι θα κάνετε για τον καταναλωτή τότε. Και μια ερώτηση, αν μπορώ να θέσω μια ερώτηση ε, για την Κομισιόν και έθεσα ε, ε, προηγουμένως κάποιος ομιλητής και η κυρία Μαγκίνες. Η αλλαγές που γίνονται τώρα στον κανονισμό για τα λοιπάσματα. Τι ακριβώς βλέπει η Κομισιόν ως έναν τρόπο να βελτιωθεί ε, ουσιαστικά η χρήση ανορόβιας δεξαμενής χώνευσης και κάποια στιγμή υπόθηκε ότι θα έπρεπε να ε, σταματήσει αυτή η ανεροβία δεξαμενή χώνευση, ε, γιατί ουσιαστικά θα μπορούσαν να σκορπιστούν τα πόβλητα. Τι πιστεύει η Κομισιόν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Σύντομη ερώτηση. Με 30 χιλιοστά βροχόπτωση πόσα, πόσα χρειάζεστε για, την, για το σύστημά σας και από πού βρίσκεται το υπόλοιπο νερό που χρειάζεστε για την στάγδιν άρδευση. Όντως τα συστήματα αυτά είναι καλά για το μέλλον. Βέβαια, οι γεωργοί έξω ρωτούν τι γίνεται με το πόση δουλειά χρειάζεται. Ενώ τον άλλο μιλτή αγροδασοκομεία. Ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν στην γερμανική γεωργία τέτοια προβλήματα. Τι απαντώ τότε σε αυτούς για να ενταχθούν τα πράγματα αυτά στα σημερινά συστήματα της αγροτικής οικονομίας. Τα συστήματα είναι πολύ αποτελεσματικά και οικολογικά ανεκτά ιδίως σε χώρες ε, του νότιου ημισφαιρίου. Μιλήσατε για το φοινικό λαδό. Θεωρείτε και τέτοια συστήματα ε, ότι προσφέρουν μια βιωσιμότητα, δηλαδή όπου ε, παράγεται το φοινικό λαδό με τους τρόπους που παράγεται. Ευχαριστώ. Είστε ο τελευταίος ερωτών. Θα δώσω πάλι το λόγο. Γνωρίζετε τώρα τους κανόνες, 3-4 λεπτά το πολύ για τις απαντήσεις σας. Εσείς πρώτος κύριε Αρπάζ για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής μας. Ως καθηγητής του Πανεπιστημίου θα μπορούσα να σας πω ότι για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας χρειάζομαι ένα ολόκληρο εξάμεινο αλλά θα προσπαθήσω. Μία από τις ερωτήσεις που κάνατε είναι πώς ε, διαδίδουμε τις πληροφορίες στους ε, γεωργούς μας. Μέσω των υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα μας, αντιλαμβάνομαι ότι το σύστημα, παρόμοιο σύστημα που υπήρχε στην Ευρώπη, extension service, δεν ε, καταργείται πλέον, ενώ το σύστημα αυτό εξυπηρετεί να διοχετεύονται οι πληροφορίες από τους επιστήμονες κατευθείαν στους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά τους νέους, όντως ανησυχούμε για το χαμηλό ποσοστό των νέων μας που μπαίνουν στη γεωργία, διότι ο μέσος όρος των Ισραηλινών γεωργών φτάνει τα 60 χρόνια. Τα ίδια που συμβαίνουν και εδώ στην Ευρώπη. Ένας τρόπος είναι χρησιμοποιώντας αυτά τα ευφυή τηλέφωνα. Δηλαδή να τους πρόξουμε να δουλέψουν πάνω στις ιδέες για τη χρήση αυτής εδώ της τεχνολογίας στην γεωργία. Πολλοί γεωργοί σήμερα κυκλοφορούν με τέτοια ευφυή τηλέφωνα στις τσέπες τους και ελέγχουν ανα πάσα στιγμή την εκμετάλλευσή τους. Με ρωτήσατε από πού βρίσκουμε το νερό στην έρημο. Το Ισραήλ είναι το... είμαστε νούμερο ένα στην αφανάτωση ανά τον κόσμο. Στο παρελθόν δεν είχαμε νερό και είχαμε ε, υποστεί τα πάνδυνα εκ της ελλείψεως αυτής. Αλλά χάρη στην τεχνολογία της αφαλάτωσης, όσο υπάρχει νερό στην Μεσόγειο, νομίζω θα είμαστε ασφαλείς. Σε ό,τι αφορά την έρημο, στο παρελθόν έφτιαξε το Ισραήλ ένα αγωγό από το βορρά του Ισραήλ μέχρι την έρημο για να μπορούμε να παρέχουμε νερό. Τώρα χρησιμοποιούμε κάποιο από το νερό που υπάρχει στην έρημο, αλμυρό νερό είναι αυτό, πάλι το αφαλατώνουμε και το χρησιμοποιούμε στη γεωργία. Βέβαια χρειάζεται να είναι κανείς προσεκτικός, διότι με τη χρησιμοποίηση, με τη χρησιμοποίηση ε, ε, α, αφαλατισμένου νερού, δηλαδή στην αφαλάτωση αφαιρούνται και ορισμένα θρεπτικά συστατικά που έχει το νερό. Και γι' αυτό χρειάζεται εκ νέου ανάμειξη ή πρόσμιξη για να μην υποστούν βλάβη τα φυτά. Άλλη ερώτηση που μου κάνατε ήταν για την επιστημονική συνεργασία. Έχουμε πολλές επιστημονικές συνεργασίες με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την μεταφορά τεχνολογίας μας σε άλλα μέρη του κόσμου. Όλο και περισσότερες χώρες του κόσμου προσαρμόζονται και υιοθετούν την τεχνολογία μας. Και ευχαρίστως λέμε ότι ε, μεγάλος αριθμός Ισραηλινών εταιριών ε, δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο για να ε, προαγάγουν την στάγδιν άρδευση και άλλες μορφές αρδεύσεως που έχουμε επινοήσει. Ίσον, σε ό,τι αφορά την διατροφή των αγελάδων μας, όπως σωστά είπατε, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ερευνάς μας είναι η μακροβιωματική έρευνα της εντερικής χλωρίδας των αγελάδων. και οι τρόποι διατροφής τους. Ε, για παράδειγμα την ε, φλούδα του ροδιού για, να, ε, για τη διατροφή των αγελάδων. Αυτός ο φλοιός των ροδιών έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά αντιοξυδοτικών. Και τελειώνω με την τελευταία ερώτηση. Ένα από τα πράγματα που έχουμε κάνει είναι να προωθούμε συνεργασίες με γεωργούς ή ε, επιχειρήσεις άλλων χωρών ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες μας εκεί και να μην χρειαστεί δηλαδή να μεταφέρουμε ολόκληρο το προϊόν από το Ισραήλ στην άλλη χώρα αλλά να μπορεί να παράγεται επιτοπίως και να ξεπεράσουμε έτσι το πρόβλημα της απόστασης. Με τέτοιου είδους συνεργασίες λοιπόν ε, ε, αποκομίζουν εισόδημα οι επιχειρήσεις μας αλλά και μετριάζεται το πρόβλημα των ε, μακρινών αποστάσεων. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερε από τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ για την ακριβιά σα και την εξωτερικιά σα, Ο κύριος Βόρμς, ευχαριστώ Πρόεδρε η ερώτηση του κυρίου Μπέλντο πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους νέους. Έχουμε διάφορα παραδείγματα από διάφορες χώρες στο Μαλάου, ή την Κίνα, την Ινδονησία, όπου ο πρόσθετος πλούτος που δίνουν ε, στα χωριά τα συστήματα ε, οδηγεί στο να μην φεύγουν, να μην μεταναστεύουν πλέον οι άνθρωποι στις πόλεις, επιστρέφουν στα χωριά και βλέπουν οι νέοι ότι μπορούν ε, να κερδίσουν αρκετά χρήματα για να παντρευτούν. Έτσι λοιπόν μένουν τόπου. Αυτό λοιπόν ανήκει στην ευρύτερη συζήτηση για τη μετανάστευση. Κύριε Άγνιου, για τον ε, χρησιμοποιούμε αυτά τα δέντρα που αναφέρατε εμείς, ε, χρησιμοποιούμε ε, χιλιάδες δέντρα, ελέγχουμε διάφορα είδη και ανάλογα με το που είμαστε στον κόσμο έχουμε πολύπλοκες ε, μίξεις ε, για τις χαρουπιές. Επίσης μας ενδιαφέρει ε, και η σειραφή των γονιδιωμάτων. Παρακολουθούμε ουσιαστικά κάποιες καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί και βλέπουμε πώς μπορούν να εξημερωνθούν ε, και για τα συστήματα αγροδοσοκομείας ε, στο Βορρά. Τα μεγαλύτερα συστήματα αγροδοσοκομείας ε, στην Ευρώπη βρίσκεται στην Βόρεια Σκανδιναβία και στη Βόρεια Ρωσία, όπου έχετε εκεί και ζώα και δέντρα, ένα μείγμα που βοηθούν το ένα το άλλο. Επίσης έχουμε και στη Σκοτία τα βοσκοτόπια και χρησιμοποιούνται ζώα παρά καλλιέργειες στα συστήματα αυτά. Και τέλος, ναι, Έχουμε μια νέα τεχνολογία, ιδιαίτερα παραδοσιακή όμως στη σημερινή γεωργία για τους περισσότερους γεωργούς είναι μια νέα τεχνολογία, δεν έχουν εμπειρία και οι ε, γειτονέ τους έχουν εμπειρία, ούτε υπάρχουν σύμβουλοι και ουσιαστικά μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο αν κάνεις ένα λάθος, αλλά είναι πολλά υποσχόμενο. Κυρία Μίλλερ σε σχέση με τα κριτήρια του Λούλου είναι καλά. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, αλλά εγώ πιστεύω ε, ότι είναι μέρος του εφιάλτη. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε απλά ε, το σύστημα αφαλού που έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί από τους περισσότερους ως ένα σύστημα, ε, θα ήταν το καλύτερο. Βέβαια, εγώ εργάζομαι σε τροπικά συστήματα, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς εδώ στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση ήταν από τον κύριο Χόισλινγκ. Ναι, η περαιτέρω ε, ουσιαστικά το περαιτέρω πρόγραμμα είναι ένα θέμα γιατί θα χρειαστείτε ε, περαιτέρω εργασία και θα έχετε ε, και κάποια δέντρα και διάφορες καλλιέργειες και πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ε, πώς θα επενδύσετε, πώς θα σκεφτείτε διαφορετικά. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι περισσότεροι γεωργοί. Έτσι λοιπόν ο λόγος είναι ότι η έρευνα δεν έχει γίνει για να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές στους γεωργούς. Όσοι χαράζουν τις πολιτικές πρέπει να διασφαλίσουν ότι γίνεται η κατάλληλη έρευνα για να έχουν τελικά οι γεωργοί κάτι πιο απτό παρά το προαισθημά τους στο οποίο να βασιστούν. Τώρα η ερώτηση για το αν μπορούμε να το κάνουμε σε μεγάλη κλίμακα ε, και σε πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις διαφωνώ μαζί σας μπορεί να γίνει ε, σε μεγάλες καλλιέργειες απλώς ε, χρησιμοποιείται διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας από αυτά που έδειξα που χρησιμοποιούνται στη Γαλλία. Ναι, θα είναι ε, ουσιαστικά πιο απλό να έχουμε πιο μικρές καλλιέργειες αλλά θα είναι πιο παραγωγική, ε, θα είναι πιο παραγωγική η καλλιέργεια. Και επίσης για το φινικέλαιο, είναι βιώσιμο, είναι τώρα μία λέξη αυτή που χρησιμοποιείται πάρα πολύ όρος βιώσιμος. Δεν ξέρω τι σημαίνει πια, αλλά αυτός ο τρόπος της παραγωγής φινικέλαιου οδηγεί σε μικρότερη διάβρωση του εδάφου, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και πιθανότητα είναι πιο βιώσιμο από τη μονοκαλλιέργεια. Σας ευχαριστώ. Merci. ευχαριστούμε κύριε Βόρμς και κύριε Χαρπάς για τις πολύ ακριβείς απαντήσεις σας και ήταν συμπληρωματικές όλες αυτές οι ομιλίες που ακούσαμε γιατί με το νέους προσανατολισμούς της κοινή γεωρικής πολιτικής είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε το γεωρικό μας μοντέλο και να προσδιορίσουμε μια δημόσια πολιτική για να συμπαρασταθούμε στη γεωργία του μέλλοντος. Και πολύ χρήσιμη αυτή η δημόσια ακρόαση μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις ε, εύστοχες ε, ομιλίες σας, ε, τις οξυδερικές απαντήσεις σας και ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Λόγκο. Προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ την κυρία Ρελή Τρουβέ να έρθει στο βήμα. Για να περάσουμε στο σημείο 5 της ημέρης της διάταξης. Την παρουσίαση της μελέτης με θέμα μέτρα κατά της ανισορροπίας στην αγορά. Ποιες είναι οι προοπτικές του ευρωπαϊκού γαλακτοκομικού τομέα μετά τις ποσοστώσεις γάλακτος. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία Εγώ είχα επιστήσει την προσοχή των συντονιστών ε, σε προηγούμενη συνεδρίαση στη μελέτη που ανέθεσε το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας σε μια διεθνή ομάδα ερευνητών από τον Καναδά, Γαλλία, κατοχώρες και η κυρία Τρουβέ είχε την καλοσύνη να μας παρουσιάσει τα πορίσματα αυτής της μελέτης γιατί ήταν η συντονίστρια αυτής της μελέτης. Ευχαριστώ ε, την ε, καλεσμένη μας που είναι καθηγήτρια ε, και μάλιστα συντονίστρια στη συγκεκριμένη μελέτη. Θα ήθελα να σας δώσω μόνο δυστυχώς ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσετε την μελέτη σας και θα ακολουθήσει η συζήτηση πριν ή μετά την παρουσίαση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Χάπς της Γενικής Διεύθυνσης Αγκρή ε, θα λάβει το λόγο μάλλον αμέσως μετά την παρουσίαση της έκθεσης και πριν τη συζήτηση με τους Ευρωβουλευτές. Αυτά και περιμένουμε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα σας μάλλον και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπατε ήμουν η συντονίστρια αυτής της μελέτης που έγινε με συνεργασία ερευνητών από τον Καναδά, τις κατοχώρες και τη Γερμανία. Δημοσιεύθηκε πριν από λίγους μήνες και το περιεχόμενό της ε, θα το βρείτε στην, ε, στο του Γαλλικού Υπουργείου Γεωργίας. Βλέπετε τον, ε, το link και θα σας κάνω μια σύνοψη αυτής της μελέτης. η μελέτη ήταν περίπου 300 σελίδες, ε, η σύνοψη περίπου 20 σελίδες. Καταρχήν, η μελέτη έγινε μέσα σε ένα χρόνο με βάση και τη βιβλιογραφία αλλά και στατιστικά στοιχεία και δημοσιονομικά στοιχεία αλλά και από συζητήσεις και συνομιλίες που έγιναν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε μελέτη και σε με μελέτες που έγιναν στον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, την ε, Ελβετία και πολλές γαλακτοπαραγωγές χώρες. Καταρχήν, είχαμε πρόσφατα μεγάλη ανισορροπία των γαλακτοκομικών αγορών και μια πτώση των τιμών από το 2014. Βλέπετε στον πίνακα αυτό το νέο πλαίσιο μεγάλης αστάθειας και διακύμαση των τιμών μετά τη μείωση ε, ε, των τιμών εγγύησεων στα επίπεδα 2005-2006. Ε, αρχικά είχαμε μία σταθερότητα τιμών, βλέπετε στη Γαλλία, η οποία έχει υπονομευθεί μετά τη δραστική μείωση των τιμών εγγύησης στις τιμές παραγωγού. Και μάλιστα σήμερα έχουμε μια χαοτική κατάσταση στις αγορές λόγω της μεγάλης αυτής αστάθειας των τιμών. Η βασική μας ανάλυση αφορούσε τα ευρωπαϊκά μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την το πέρας των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Είχαμε μια διαρθρωτική πλονοσματική παραγωγή με υπερτίμηση βέβαια της παραγωγής και μετά τη μείωση των τιμών είχαμε ισχυρή αύξηση της παραγωγής. Και μάλιστα το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που συνέβαλε το περισσότερο στην πλανοσματική παραγωγή παγκοσμίω. Συνέβαλε έτσι στην περαιτέρω μείωση των τιμών. Δεν ήταν η πρώτη πλανοσματική ε, παραγωγή αυτή των Ηνωμένων Πολιτών της Νέας Ζηλανδίας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εφοδίαζε τις παγκόσμιες αγορές με πλεονασματική παραγωγή γάλακτος. Και επίσης υπερτιμήθηκαν και η διέξοδοι και εξαιτίας της ίσω ίσως και της ε, ζήτησης ε, της Κίνας αλλά και του ρωσικού εμπάργου. Επίσης, ε, τη στιγμή που λήφθη η απόφαση για την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, δεν έλειψαν υπόψη οι συνέπειες που θα είχε αυτή η περάτωση των ποσοστώσεων στην μείωση του ιωρικού εισοδήματος και στη διάβρωση της επενδυτικής τους ικανότητας που μάλιστα δεν ε, κράτησε μόνο ένα χώρο, είχαμε μια γεωγραφική κατανομή αυτών των ε, προβλημάτων. Και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ε, έχουμε την έννοια της κρίσης, αλλά της ατέλειας των αγορών περισσότερο. Και μάλιστα με εργαλεία που κατά τη γνώμη μας διαχειρίζονται εκ των υστέρων την αστάθεια των τιμών, τη μεγάλη διακύμαση αυτών των τιμών και δράζονται κυρίως σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Και μάλιστα η ιδιωτική αποθεματοποίηση, η, μάλιστα, δημόσια αποθεματοποίηση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και μάλιστα 220 ε, ευρώ τόνος είναι η τιμή παρέμβασης ε, και μάλιστα είναι τελείως αναποτελεσματική αυτή η τιμή και το είδαμε πριν στον πίνακα με τις εξελίξεις των τιμών. Αυτή η χαμηλή τιμή δεν συμβάλλει στη σταθεροποίηση και μάλιστα εξαιτία περίοδου ενεργοποίηση το 2014 ήταν τελείω αναποτελεσματική η χρήση αυτή τη τιμή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ιδιωτική αποθεματοποίηση, στην οικονομική βιβλιογραφία έχουμε πολύ μεγάλους περιορισμούς της ιδιωτικής αποθεματοποίησης με τον κίνδυνο ε, να μην έχουμε μετάβαση των των τιμών στον παραγωγό ή κερδοσκοπικές ε, ενέργειες με απροσδόκητα αποτελέσματα. Επίσης, ε, είχαμε την πρώτη διετία μεγάλη ανισορροπία της αγοράς και τα μέτρα ε, παρέμβασης της αγοράς ήταν αναποτελεσματικά. Και μάλιστα το άρθρο 222, που είναι το άρθρο που ισχύει από τότε που προβλέπει η θελοντική μείωση της παραγωγής σε αντάλλαγμα κάποιες άμεσες ενισχύσεις. Ναι, μεν, το άρθρο αυτό συνέβαλε σε μια μείωση της παραγωγής ή τουλάχιστον σε μια ακαλμία σε ό,τι αφορά την αύξηση της παραγωγής σε μερικές χώρες και δει την Γερμανία και τη Γαλλία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά αυτό το άρθρο δεν, ε- δεν οδήγησε σε μείωση της παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι κατοχώρες Ιρλανδία ή το Βέλγιο συνέχισαν να αυξάνουν την παραγωγή τους. Ε, για παράδειγμα, δεύτερο εξάμεινο ε, είχαμε αύξηση 7% στι κατοχώρε. Επίσης, το άρθρο 226 που μιλάει για το αποθεματικό της κρίσης ε, δεν εφοδιάζεται με αρκετά κονδύλια αυτό το αποθεματικό και από την αρχή της κάθε εξαντλείται λόγω του χαμηλού επίπεδου. Επίσης έχουμε κάποια μέσα ε, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωρικής πολιτικής, ε, κάποια ταμεία αμοιβαιοποίησης. Ε, στον πρώτο πυλώνα είχαμε την κοινή οργάνωση αγοράς, στο δεύτερο πυλώνα έχουμε την εφαρμογή των ταμείων αμοιβεοποίησης μόνο σε τρία σχέδια ανάπτυξη πέθρου και μάλιστα η χρήση των ταμείων αμοιβεοποίησης είναι πολύ περιορισμένη εξαιτίας των απαιτήσεων του ΠΟΕ και κάποιων δυνατοτήτων που δεν αξιοποιούνται. Τέλος, είχαμε και το παρατηρητήριο της ε, γαλακτοκομικής αγοράς, ε, πολύ θετική παρουσία του παρατηρητηρίου, αλλά ε, είναι λίγα τα στοιχεία που συγκεντρώνουν σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επίση, το άρθρο 221. Το άρθρο τη κοινή Οργάνωση αγορά, του πρώτου πυλώνα που επιτρέπει ακόμη περισσότερες δράσεις για, το, για τον υποχρεωτικό περιορισμό της παραγωγής που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Έχουμε μέτρα που δεν είναι αρκετά φιλόδοξα όμως και δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τη διαρθρωτική κρίση της πλεονασματικής παραγωγής. Επίσης τώρα να συγκρίνω την εφαρμογή σε διάφορες χώρες μέλη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στην παραγωγή και για τη συμμετοχή των συνεταιρισμών στη μεταποίηση. Σε ορισμένες περιοχές πάντως έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση του κλάδου γιατί μερικές φορές ε, στις κατοχώρες, στην Ιρλανδία ή στη Δανία έχουμε σχεδόν μονοπόλιο των συνεταιρισμών, αλλά σε άλλες χώρες και σε άλλες ε, περιφέρειες ε, έχουμε ιδιωτική και μετα... Ε, βιομηχανίες ε, ε, και όχι μεγάλη ενεργοποίηση των συνεταιρισμών. Στη Νότια Γερμανία έχουμε πιο ιστορική οργάνωση παραγωγών, αλλά στη Γαλλία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε σύναψη συμβολέων με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής και τα εργοστάσια με ένα πολύ αρνητικό απολογισμό δεν είναι μεγάλη η σχέση των συνεταιρισμών και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική επανισορρόπηση των ε, δυνάμεων του κλάδου, δηλαδή των παραγωγών απέναντι στα αργοστάσια μεταπίεσης. Επίσης, σε ορισμένες περιοχές έχουμε μεγάλη γαλακτοκομική πυκνότητα και το 2015-2016 στην Ιρλανδία και στις κάτω χώρες ε, είχαμε μεγάλη αύξηση της παραγωγής ε, το σχέδιο της, Γερμανίας, της Ιρλανδίας για το 2020 και θεωρούσαν ως εναλλακτικό πρόγραμμα σε σχέση με το, με το πέρας των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, αλλά σε άλλες περιοχές ε, δεν είχαμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η Ιρλανδία λόγω της πλονεσματικής παραγωγής και είχαμε μείωση τελικά της παραγωγής. Έχουμε μεγάλες ανισότητες ε, και ως προς την παραγωγή και ως προς τη γεωγραφική κατανομή. Επίσης, ακόμη και στις περιοχές που αυξάνουν την παραγωγή τους και εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για τους γαλακτοπαραγωγούς. Ακόμη και στην Ιρλανδία, στη Γερμανία και τις κάτω χώρες. Με αρνητικό σχετι... συσχετισμό δυνάμεων απέναντι στους μεταποιητές όταν δεν είναι αυτοί οι συνεταιρισμοί και μια, ένα σχετισμό δυνάμεων που αποβαίνει εις βάρος των παραγωγών. Επίσης, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες περιοχές, Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδάς, ε, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Έχουμε δύο άκρε. Στη Νέα Ζηλανδία δεν έχουμε σχεδόν καμία ρύθμιση τη αγορά, αλλά μονοπόλιο στην εξαγωγή της ε, εταιρεία Φοντέρα. Ενώ στο άλλο άκρο έχουμε τον Καναδά, που έχει τις ποσοστώσεις, ε, υψηλούς δασμούς, τιμές παρέμβασης και τα έχει κρατήσει αυτά όλα στην εσωτερική αγορά. Η, η Νέα Ζηλανδία έχει απορριθμίσει τα πάντα και είναι εξωστρεφής, αντίθεση με τον Καναδά που είναι εσωστρεφή με μεγάλη ρυθμίση της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ των δύο ακραίων μοντέλων έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε και, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και την Ελβετία με ένα ιδιόρυθμο σύστημα έχουν περίπου 2.500 ευρώ το εκτάριο άμεση ενίσχυση στο γαλακτοπαραγωγό στην Ελβετία. Ένα τελείω ιδιαίτερο σύστημα. Εμείς έχουμε 300 ευρώ το εκτάριο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 2.500 ευρώ ανά εκτάριο στην Ελβετία. Βλέπετε τεράστια διαφορά στις επιδοτήσεις. Τώρα, στις Ηνωμένε Πολιτείες... Δεν έχουν μόνο δημόσιες ενισχύσεις ασφαλιστικού χαρακτήρα, δηλαδή ε, παίρνει κανείς μια δημόσια ασφάλιση με διάφορες επιλογές και ανάλογα με την κάλυψη που θέλει, όσο μεγαλύτερη κάλυψη θέλει, τόσο υψηλότερο είναι το ασφάλιστρο, αλλά δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό το σύστημα, γι' αυτό και οι περισσότεροι παραγωγοί προτιμούν την ε, χαμηλότερη κάλυψη, που από το 2014 δεν έχει ενεργοποιηθεί από τη μείωση των τιμών και μετά. Οπότε στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σημαντικό σύστημα στήριξη, όχι μόνο μέσω των δημόσιων ενισχύσεων, αλλά κυρίω μέσω του συστήματο καθορισμού των τιμών, του Mixed Marketing Orders. Έτσι, ανά πολιτεία ή ανά ομάδες πολιτιών έχουμε καθορισμό της τιμής ε, του γάλακτος ανά τμήμα αγορά. Υπάρχει ξεχωριστή τιμή για τον απογάλα για το γιαούρτι, το τυρί και επίσης οι ε, διακλαδικές οργανώσεις έχουν μία τιμή για όλους τους παραγωγούς της πολιτείας και όλοι οι παραγωγοί λαμβάνουν την ίδια επιδότηση. Και στη συνέχεια οι μεταποιητές καταβάλουν την, ε, την τιμή του γάλακτος ανάλογα με το τμήμα της αγοράς και την ποιότητα του γάλακτος. Το ίδιο ισχύει και στον Καναδά. Και στην Ελβετία έχουμε ένα σύστημα διάκριση των τιμών σε ε, επίπεδο Ελβετίας με βάση τα τμήματα της αγοράς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις χώρες που δεν έχουν συνεταιριστικό μονοπόλιο αφήνουμε τους ε, μεμονωμένους ε, οι ή μικρές ομάδες παραγωγών και η λήψη της δημόσιας ε, ρύθμιση, του αφήνουμε να διαπραγματευτούν μόνοι του τις συνθήκες απέναντι σε μεγάλες εταιρείε μεταπίεση. Είναι ανευπροηγουμένο αυτή η κατάσταση αν συγκρίνουμε τι ισχύει σε άλλους μεγάλους παραγωγούς. Ακόμη και στην ε, ε, Νέα Ζηλανδία όλοι οι παραγωγοί λαμβάνουν την ίδια τιμή γιατί η Φοντέρα έχει το μονοπόλιο τη εξαγωγή. Και οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι στο τέλος του έτους λαμβάνουν τα μερίσματα, οπότε έχουν μια επιστροφή προς το τέλος του έτους η γαλακτοπαραγωγή. Η ομάδα των ερευνητών ε, που εκπώνησε τη μελέτη θεωρεί ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να διέλθουμε από αυτή τη διαρθρωτική κρίση της παραγωγής χωρίς να έχουμε υποχρεωτικό μηχανισμό ελέγχου της παραγωγής σε περίπτωση κρίσης. Γιατί βλέπουμε σήμερα που είναι θελοντική η μείωση της παραγωγής ότι δεν ε, έχουμε συνολική μείωση της παραγωγής ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε υψηλότερε τιμές γάλακτος. Σήμερα η μείωση των τιμών, η πτώση των τιμών συνεχίζεται. Και ε, το μέλλον είναι αβέβαιο. Και το γεγονό ότι άλλε χώρε συνεχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή του, άλλε περιοχέ συνεχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή του, δεν μα επιτρέπουν να επιστρέψουμε σε υψηλότερες τιμές. Ε, χρειάζονται μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση της υπερπαραγωγής. Εμείς έχουμε ένα σύστημα κυρώσεων για την ε, υπερπαραγωγή σε περίπτωση κρίσης, υποχρέωση είτε διατήρησης είτε μείωσης της παραγωγής σε περίπτωση κρίσης και παράλληλα ενισχύσεις για τη μείωση της παραγωγής. Άλλες δυνατότητες θα ήταν ε, να περιορίσουμε κάποιους μηχανισμούς στήριξης ε, ε, για αυτούς που μειώνουν την παραγωγή τους. Το Ολλανδικό Σύστημα Ποσοστώσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα και τέλος θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιους συμπληρωματικούς μηχανισμούς ε, για το εισόδημα σε περίπτωση κρίσης ή μέσω κάποιων ταμείων αμοιβιοποίησης ή με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Αποθεματικού ε, Κρίσεων ή κάποιες αντισυγκυριακές πληρωμές. Γιατί δεν έχουμε ένα πραγματικό μηχανισμό συμπλήρωσης του εισοδήματο που θα, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις των τιμών. Επίσης έχουμε κάποιες ε, πολύ πιο ε, ευάλωτες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή περιοχές με δυσμενείς συνθήκες. αυτός θα πρέπει να καλυφθούν από τον πρώτο πυλώνα ή να προβλέψουμε καλύτερη κατανομή των κυκλωμάτων διανομής. Και ίσως και μια πραγματική επισητιστική πολιτική για την ΚΑΠ μετά το 2020. Και επίσης να διαφυλάξουμε τις ε, δασμολογικές, ε, τους, ε, τους δασμούς, που είναι η τελευταία ασφαλιστική δικλίδα, τουλάχιστον για τα καλοπτοκομικά προϊόντα. Οπότε προσοχή με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχετε ασχοληθεί εδώ και πολύ καιρό. Μπράβο σας. Λοιπόν, θα δώσω κατευθείαν ε, το λόγο στην Κομισιόν. Στον κύριο Σάψη θα του ζητήσω να είναι βέβαια σύντομος στην παρέμβασή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, κυρία Τρουβέ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ε, εξετάσαμε εξ του συνεγγύης ε, όχι μόνο την περίληψη αλλά και την ίδια την έκθεση. Και πράγματι πρόκειται για μια πολύ πλούσια και ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης στις διάφορες χώρες στο γαλακτοκομικό τομέα. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πρέπει όμως να παραδεκτώ ότι κάποια από τα συμπερίσματά σας που προκύπτουν από αυτή τη βασική ανάλυση δεν μας βρίσκουν 100% ε, σύμφωνους, δηλαδή τους δικούς μας αναλυτές. Τώρα, για να περάσω απευθεία ε, στα συμπεράσματα και στις ε, συστάσεις ε, που κάνατε στην έκθεση. Νομίζω ότι η κύρια σύσταση είναι η πρώτη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι συστάσεις είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αποφάσισαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πριν δύο χρόνια περίπου για να ε, επιλύσουν ε, το πρόβλημα στο γαλακτοκομικό τομέα και για να παράσχουν ε, το απαραίτητο πεδίο εφαρμογή για έναν ανταγωνιστικό γαλακτοκομικό τομέα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν 11 άλλες συστάσεις που είναι εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες και θα έκανα εδώ ένα σύνδεσμο με αυτά που συζητήθηκαν πρόσφατα και στο Συμβούλιο Γεωργίας την έκθεση Βέρμαν, όπως αποκαλείται. Ήταν το αποτέλεσμα της ε, μελέτης ε, που έκανε η Task Force για τη Γεωργία τους τελευταίους εννέα μήνες. Και πολλές από τις δευτερεύουσες συστάσεις ε, που έχετε υποβάλει στην έκθεσή σας ανήκουν και στη δεσμή που παρουσίασε η ομάδα Βέρμαν. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε πολλούς κοινούς τόπους και μπορούμε φυσικά να αναπτύξουμε ιδέες και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, λιγότερο ευνοούμενες περιοχές και τις περιοχές ε, σε ό,τι αφορά την τοπική παραγωγή αλλά και, ε, και τον επισητισμό υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρεται εκεί για τη διαφάνεια για το πώς θα οργανώσουμε την ε, κυκλοφορία των πληροφοριών στην αγορά για όσους χρειάζονται περισσότερο διαφανείς πληροφορίες. Και επίσης έχουμε και το μεγάλο μέρος της ε, σύναψης συμβάσεων και της ε, μαζικής προσφοράς. Υπάρχουν εδώ διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν δημοσίως, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει τα τελευταία δύο χρόνια και είμαι σίγουρος ότι Υπάρχει πεδίο εφαρμογή, ε, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εκτός ε, από την πρώτη σύσταση. Όπως ξέρετε και η Κομισιόν αλλά και το Συμβούλιο που συζητούν αυτό το θέμα ξέρουν ότι χρειαζόμαστε αλλαγή στο βασικό κανονισμό. Επομένως ε, είναι θέμα του συνομοθετών να αλλάξουν εντελώ αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ε, τεράστια δουλειά, για το πολύ μεγάλο έργο σας και θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Θα σας δώσουμε χρόνο για τις απαντήσεις στη συνέχεια. Να δώσουμε τώρα τη συζήτηση στους βουλευτές. Ένα λεπτό ο καθένας ε, έχετε για την παρέμβασή σας. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Λουαζό. Να ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τρουβέ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ε, δηλαδή τι γίνεται μετά το τέλος ε, των ε, ποσοστώσεων. Είναι δραματικές οι προπτικές κυρίως για όσους επιδίδονται σε παραδοσιακή γεωργία και όχι σε βιομηχανική γεωργία και αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γαλλική Ομοσπονδία των Γαλακτοπογών προβλέπει ότι θα εξφανιστούν 10.000 γαλακτοφόρες ε, ε, αγελάδες και ο υπουργό Γεωργίας μας ε, ουσιαστικά πύχησε τις προτάσεις του Ελεύθερου Συνδικάτου και πρότεινε να υπάρχει αλλαγή του επαγγέλματος των γεωργών και μετατροπή και επίσης εκτιμάται ότι θα δούμε στην πραγματικότητα συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων και όχι μείωση ε, της παραγωγής. Έχουμε μία μελέτη που λέγεται μέτρα κατά της ανεπερισορροπίας στην αγορά, ποιες προοπτικές ε, για ε, τις ποσοστώσεις στη ζάχαρη στον τομέα στον ευρωπαϊκό τομέα της ζάχαρης. Η Κομισιόν γνωρίζει ε, ουσιαστικά την, για το πώς η αναταραχή φέρνει στο γεωργικό τομέα. Ευχαριστώ. Κύριος Ντές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ανάπτυξη του θέματος από την κυρία Τρουβέ. Έχω ορισμένα σχόλια. Μόλις πριν ακούσαμε για ποσότητες βουτύρου, 30.000 προτείνει η Κομισιόν, να αφαιρεθούν από την αγορά. Άλλοι μίλησαν για 250.000 τόνους. Βλέπετε τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι τιμές, να σταθεροποιηθούν τουλάχιστον με την αφαίρεση αυτών των ποσοτήτων. Μέσα σε τρεις μήνες, ωστόσο, η τιμή ανήλθε η μεγαλύτερη αύξηση τιμής η μεγαλύτερη αύξηση τιμής εδώ και 20 χρόνια. Καλά θα ήταν να υπήρχε ωστόσο κάποια αποθήκευση ε, ποσοτήτων βουτύρου για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί πάλι προς τα κάτω η τιμή. Γι' αυτό είναι, αυτή, αυτό το νόημα της ερώτησή μου. Μήπως πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί καλύτερα ώστε να αποκατασταθεί κάποια σταθερότητα στην αγορά. Ευχαριστώ κύριε Ρομπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ομιλήτρια η οποία αναφέρθηκε στους κύριους λόγους για τους οποίους προέκυψε η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. και αν ήταν πάλι οι τιμέ του τελευταίους μήνε. Έχει βελτιωθεί λοιπόν κάπως η κατάσταση. Το μέλλον είναι ακόμα άδειλον. Μπορεί να ακολουθήσει και άλλη κρίση μέσα σε έξι μήνες και ίσως και χειρότερη. Είναι αλήθεια ότι το ρωσικό εμπάργκο έχει βαρύτατες επιπτώσεις σε χώρες όπως η Λιθουανία και οι άλλες βαλτικές χώρες. Οι Ρώσοι ωστόσο εξακολουθούν να καταναλώνουν γάλα και δεν έχει μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση. Άρα κάτι λάθος υπάρχει εδώ. Και δεν μπορούμε να έχουμε καμιά ασφάλεια στις μελλοντικέ πρόπτικες. Στο πρώτο μέρος της σημερινής συνεδρίασης μιλήσαμε, ε, αναρωτηθήκαμε για τους λόγους που οι νέοι άνθρωποι δεν εισέρχονται στη Γεωργία, διότι δεν βλέπουν μέλλον στη Γεωργία. Αυτός είναι ο λόγος. Και πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών θα ταχθεί υπέρ ενό υποχρεωτικού μηχανισμού. Κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναζητηθούν τρόποι. Ευχαριστώ, κύριο Χόισλινγκ. Πολύ ενδιαφέρον βρήκα ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως κατανοεί στο τέλο ότι αυτή η απελευθέρωση τη αγορά δεν ήταν το καλύτερο μέσον. Εσείς μελετήσατε διάφορες αγορές και μάλιστα και αγορές ιδιαίτερα αυστηρά ρυθμισμένες όπως του Καναδά που βλέπουμε τώρα και με την ΣΕΤΑ. Τι γίνεται εκεί, ποια είναι εκεί η κατάσταση. Είπατε προς το τέλος της ομιλίας σας ότι θα έπρεπε να καθοριστούν υποχρεωτικά κάποια ποσοστά, κάποιες ποσότητες παραγωγής. Ε, τότε πώς θα το λέτε αυτό αν δεν το λέτε ποσοστώσεις. Κάποιοι άλλοι λένε εδώ ότι για την ώρα ανέρχονται οι τιμές. Ναι, αλλά σε ποιο επίπεδο. Και ε, διαρωτώ με, εάν οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ισοσταθμίσουν τις απώλειες που είχαν τα τελευταία χρόνια, θα ξαναφτάσουμε σε δύο χρόνια πάλι στα ίδια. Υπερβολική παραγωγή, μειωμένη ζήτηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι όλο αυτό το γάλα και πρέπει κάποιος να το αναγνωρίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική του ότι Πολύ μόνο και περισσότερο γάλα και ότι αυξάνει σε αριθμού η, μεσ... η, μεσαία τάξη και αυτή θα αγοράζει όλο και περισσότερο, τελικώ δεν αποδεικνύεται αληθή. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία για αυτή την ε, μελέτη. Καταρχήν ε, θα ήθελα να χαιρετήσω αυτό που αναφερθήκατε. Ε, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το θέμα, κυρίως στη Βόρεια Πορτογαλία και πρόκειται ουσιαστικά για ανισορροπία και ο κλάδος πάντοτε ζημιώνεται. Εγώ θέλω να σας πω ότι ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε συστήματα προστασίας των καταναλωτών όταν έχουμε μηνύματα ε, ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε την τιμή που πληρώνεται στους γεωργούς ε, και θέλω να αφερθώ σε τρία συγκεκριμένα μεταπροστασίας ε, του να καθοριστούν ε, οι τιμές, όπως παραδείγματο γίνεται στις Ηνωμένες Μπορείτε να μας πείτε πώς θα μπορούσε να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και υποχρεώσεις ρύθμισης της παραγωγής στην περίπτωση κρίσης και τη μέτρα συμπλήρωσης εισοδήματος ε, στην περίπτωση κρίσης. Η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη αυτοί οι τρεις μηχανισμοί θα πρέπει να ειδωθούν ε, με ανεξάρτητο τρόπο ή με διαρθρωμένο τρόπο και ε, σε ποιο βαθμό ουσιαστικά θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, είτε ο καθένας ξεχωριστά στο σύνολό τους. Ευχαριστώ κυρία Όκους. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα μελέτη. Πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε ο τρόπο με τον οποίο συγκρίνατε διάφορες χώρες όπως Καναδά, Νέα Ζηλανδία κλπ. Εγώ θα ήθελα να είχατε περιλάβει και την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει επίσης μια πολύ προστατευμένη αγορά και μια παραγωγή η οποία κατευθύνεται στην εσωτερική της αγορά. Και εκεί απολαμβάνουν οι γεωργοί πολύ σταθερέ τιμέ, όπω και στον Καναδά. Ενδιαφέρον είναι και η περίπτωση τη νέα Ζηλανδία θεωρούμε πάντοτε ότι μέσω των συνεταιρισμών μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά στην Νέα Ζηλανδία υπάρχει μόνο ένα συνεταιρισμό και επομένω δεν έχει απολύτω κανένα ανταγωνισμό. Αλλά ούτε έτσι λύνεται το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τον αγορά, δηλαδή να παρέμβουμε ρυθμιστικά στην αγορά, τουλάχιστον όταν βλέπουμε ότι πάει να ξεφύγει. Και βεβαίω όχι να περιμένουμε να ξεφύγει πρώτα, διότι είναι πολύ δαπανηρή υπόθεση αυτή όταν πια οι εκμεταλλεύσεις έχουν χάσει πολλά χρήματα και οι ζημιές ανέχονται σε 3,2 δισεκατομμύρια στη Γερμανία κάθε χρόνο και ε, υποχρεώθηκαν να, ε, να αντιμετωπίσουν τέτοιου ζημίες τον τελευταίο χρόνο. Έτσι δεν μπορεί να συνεχίσουν στο μέλλον. Ο κ. Φλάνναγκαν, ευχαριστώ. Μιλήσατε για την αγορά τη Νέα Ζηλανδίας και για την καναδική αγορά. Μιλήσατε επίση για την καναδική αγορά και είπατε ότι είναι σχεδόν το ίδιο αυστηρά ρυθμισμένε και επιδοτούμενες. Διερωτώ με εν ώψη τη πέμπτη συστάσεώ σα, τι λέτε για την πρόταση της ΣΕΤΑ. Ο Καναδάς ρυθμίζει και επιδοτεί περισσότερο. Τι επίπτωση θα έχει λοιπόν η ΣΕΤΑ εν ώψη αυτού του γεγονότο. Ε, κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ. Και η Κροατία ως νέα χώρα μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπέστη και αυτή την κρίση και τετραπλασιάστηκε ε, η εισαγωγή γάλακτος από το 2012 μέχρι το 2014 και χρεοκόπησαν 3.500 γαλακτοπαραγωγοί. Ε, Εξαιτία της κρίσης στο γαλακτοκομικό τομέα, το τελευταίο χρόνο 2.000 ε, οικογένειες ε, έχασαν την απασχόλησή τους και τον βιοπορισμό τους. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε αυτή την κρίση, γιατί συνεχίζονται οι χρεοκοπίες των γαλακτοπαραγωγών και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα χρεοκόπησαν φέτος 200 παραγωγή. Μας κάνατε κάποιες συστάσεις, πέραν των συστάσεων. Ε, θεωρείτε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ παλιών και νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την κατάσταση ε, στην παραγωγή γάλακτος μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών, βορείων και νοτίων. Μήπως θα πρέπει να έχετε ειδικέ συστάσεις αναχώρα ανάλογα με τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ. εγώ και η Μαριάννα Πεντήρ καταγόμαστε από γειτονικέ χώρες, οπότε έχουμε παρόμοια προβλήματα. Και εγώ παρόμοιους προβληματισμούς και ερωτήσεις έχω. Η κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και άλλες ε, περιστάσεις επηρέασαν την αγορά γάλακτος και δημιούργησαν τεράστια ανισορροπία. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ ε, τη Ανατολική Ευρώπη των Βαλτικών χωρών και των Δυτικών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανώσει των παραγωγών είναι διαφορετικές, η οργάνωση των παραγωγών και η ιδιοκτησία. Ε, γιατί στη Σλοβενία η μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία είναι η Λακτάρη. Και είδαμε η τιμή ε, να έχει πέσει από 35 σε 25 λεπτά και σήμερα έχει αυξηθεί κατά ένα λεπτό μόνο. Ε, βρισκόμαστε σε μεγάλη κρίση και σίγουρα δεν ισχύει θεμητό εμπόριο, δίκαιο εμπόριο, fair trade στο γάλα. Μιλάμε για fair trade με την Αφρική, γιατί δεν μιλάμε για fair trade ε, στο εμπόριο γάλακτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη σας, ε, οι μακροπρόθεσμες λύσεις τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν, ε, ρυθμισμένη παραγωγή, επαναφορά των ποσοστώσεων, οικειοθελή, εθελοντική μείωση της παραγωγής. Η πείρα σας, τι σας ε, οδηγεί ως καλύτερη λύση, πρόταση για καλύτερη λύση ή θέλουμε, θα πρέπει να επιδιώξουμε καλύτερη οργάνωση των συνεταιρισμών και των παραγωγών γάλακτος. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Κύριο Σάγνιου. Ευχαριστώ. Μιλούσαμε για κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα και τώρα ας μιλήσουμε για μια κρίση ε, για την ε, πουτίγκα γιατί δεν έχουμε αρκετό βούτυρο για την κρέμα στη Βρετανία και χρειάζεται χρόνος για να ξαναπαράγουν οι αγελάδες. Μπορεί να χρειάζονται τρία χρόνια ενώ όταν να σταματήσει η παραγωγή είναι εύκολο. Σκοτώνεις αγελάδες ενώ την ξαναρχίσεις είναι δύσκολο για να δούμε. Ε, θα στραφούμε στην Ιρλανδία και στις κάτω για να μας βοηθήσουν να καλύψουμε αυτό το κενό. Έτσι λοιπόν, ε, ποιος ε, είπε ότι το Brexit ε, δεν ήταν bad business, αλλά... Για να σοβαρέψω, φαίνεται ότι πολλοί είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος για το γαλακτοκομικό τομέα. Ε, υπάρχουν ε, διάφοροι παράγοντες που πρέπει να συντονιστούν ε, μεταξύ των διαφορών κρατών μελών και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. θέλετε να μιλήσω ένα λεπτό, θα συνεργαστώ γι' αυτό πρόεδρε γιατί θα μπορούσα να συνεχίσω και να πω πολλά. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνης. Πρόεδρε, γίνεται <laughs> κάπως συνήθεια να μιλώ μετά τον κύριο Άγνιο. Τέλος πάντων είναι καλή συνήθεια. Είμαστε ικανοποιημένοι στην Ιρλανδία και ευχαρίστω εμεί στην Ιρλανδία και νομίζω και κατά χώρε ε, να μπορέσουμε ε, και μετά το Brexit αλλά να συνεχίσουμε να δίνουμε βούτυρο και κρέμα γάλακτο στη Βρετανία. Αλλά μπορείτε να μου υπενθυμίσετε τι είπατε ε, για την Ελβετία, για τι επιδοτήσει, γιατί έγραψα 2.500 ευρώ ένα εκτάριο και είπατε στην Ευρώπη είναι 300 ευρώ ένα εκτάριο. Μάλιστα, καλά άκουσα. Και δεύτερον, όταν ε, λέτε ε, μέτρα υποχρεωτικής διαχείρισης της παραγωγής, θα χρειαστεί να έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων ή κάτι ανάμεσα. Δηλαδή, η ελεύθερη παραγωγή και κάποια διαχείριση και είναι εφικτό κάτι τέτοιο, μπορούμε να το διαχειριστούμε στην πράξη. Και σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, γιατί φυσικά ε, είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων το εμπόριο. Σε κάποιες αγορές που προσπαθούμε να έχουμε πρόσβαση είναι καλό ε, να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Τρούβε. Ξέρετε και εσείς ε, τους κανόνες, πέντε λεπτά. <laughs> Θα σας δώσω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσω να μην ακρηγορήσω για να μην αργήσετε και εσείς με τη συνεδρίασή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού στις ερωτήσεις και λυπάμαι για όσους δεν θα έχω αρκετό χρόνο ή την εμπειρογνωμοσύνη. Καταρχήν, εμείς αυτό που προωθούμε στην πρώτη σύσταση είναι ακριβώ όχι μόνο ένα μηχανισμό όπω αποφασίστηκε φέτο μέσω του άρθρου 222 για την εκούσια μείωση ε, σε ό,τι αφορά ε, την ε, μείωση τη ενίσχυση για όσου μειώνουν την παραγωγή του. Αλλά εμεί θεωρούμε ότι έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια από τα που δόθηκαν γιατί καταναλώθηκε ο προπολογισμό από κάποιου παραγωγού που ήθελαν να μειώσουν την παραγωγή του σε κάποιες εβδομάδες. Όμως, θεωρούμε ότι αν αυτό δεν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να οδηγήσει σε μειώσεις παραγωγής ορισμένες περιφέρειες, αλλά και σε αυξήσει παραγωγής αλλού από την πλευρά των παραγωγών ε, που λένε «Α, να, αυτοί μειώνουν, εμείς θα αυξήσουμε γιατί ξέρουμε ότι ίσω θα διατηρηθούν οι τιμές». Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν απαντούμε στην υπερπαραγωγή της αγοράς. Γιατί είδαμε στην Ιρλανδία, στις κατοχώρες, στη Δανία, Ιρλανδία, κατοχώρες Βέλγιο, υπήρχε αύξηση της παραγωγή ε, συνολικά στο 2016 και μιλάμε για ισχυρή αύξηση. Αυτό επίσης προτίθηκε στο γαλλικό memorandum του Ισγαλίας το 2016, δηλαδή να ενεργοποιηθεί το άρθρο 221 και όχι το άρθρο 222 που επιτρέπει αυτό που αποκαλούσαμε το 2013 και θυμάμαι τη σύνθεση που κάναμε στην διάσκεψη για το μέλος του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και τη τυθενότητας ε, μια υποχρεωτική μείωση για όλου σε περίπτωση κρίση. Δηλαδή δεν μιλάμε για να ε, επιστρέψουμε στι προηγούμενε ποσοστώσεις, αλλά να υπάρχει μείωση τη παραγωγή σε περίπτωση κρίση. Μου φαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη και όλε τι περιφέρειες. Εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το μέτρο και το μόνο μέτρο που θα ήταν αποτελεσματικό σε περίπτωση κρίση υπερπαραγωγή, όπω έχουμε σήμερα. Και να δράξω την ευκαιρία για να πω το εξή. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη σε κρίση. Η τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό έχει σταθεροποιηθεί, αλλά συνεχίζει να μειώνεται σε πολλές περιοχές. Και δεν βλέπουμε αύξηση της τιμής που καταβάλλεται στον παραγωγό. Βέβαια, στις διεθνείς αγορές υπάρχουν ε, κάποια μηνύματα για το βούτυρο, αλλά όχι για τη σκόνη, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση σε σκόνη. Όμω, αν θέλετε για την τιμή που καταβάλλεται στο παραγωγό, είτε αυτή συνεχίζει να μειώνεται, είτε διατηρείται. Όμω, σε κάθε περίπτωση δεν βλέπουμε νέα άνοδο τη τιμή. Και καθώς αναφερθήκατε στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουν οι γαλοκτοπαραγωγοί στη Γαλλία, υπάρχει μια ανάλυση που μας επιτρέπει να δούμε ότι το 1 τέταρτο των γαλοκτοπαραγωγών στη Γαλλία το 2015 είχαν αρνητικό εισόδημα. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε το 1 τέταρτο των παραγωγών με αρνητικό εισόδημα και αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες με πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση του τομέα για να απαντήσω για το συνδυασμό των εργαλείων. Ναι, πρέπει να συνδέσουμε ουσιαστικά ένα εργαλείο διαχείρισης της παραγωγής σε περίπτωση κρίσης, να υπάρχει μία υποστήριξη για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος είτε ουσιαστικά με τα μία είτε θα υπάρχουν ε, αντικυκλικές πληρωμές. Αυτό θα συζητηθεί βέβαια στα πλαίσια της ΠΑΚ μετά το 2020, της ΚΑΠ μετά το 2020. Υπήρχαν και κάποιες ανησυχίες ε, που εκφράστηκαν από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, από τα νέα κρατημέλη, τι συμβαίνει με τις εκμεταλλεύσεις ε, σε περιοχές που έχουν μειονεκτήματα. Όλα αυτά νομίζουμε ότι συνδέονται. Όμως νομίζουμε ότι η σύσταση υπερθυμών 1 για τη διαχείριση των όγκων είναι κάτι απαραίτητο αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση της υπερπαραγωγής. Και για να κλείσω. για το, σε ό,τι αφορά τα άλλα κράτη και κυρίως τον Καναδά. Ναι, στον Καναδά υπάρχουν ε, ταυτόχρονα ποσοστώσεις και μία τιμή παρέμβασης ε, η οποία αριθμίζεται στο ποσοστό ανάλογα με το ποσοστό παραγωγής ανά παραγωγό και κοινά σχέδια ανά επαρχία. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που καθορίζονται από τον κλάδο και από το κράτος, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτό το σύστημα που εμεί δεν έχουμε, δηλαδή του καθορισμού των τιμών μέσω του κλάδου, υπό την εποπτεία του κράτους. Στον Καναδά έχουμε το συνολικό πακέτο. Έτσι λοιπόν, ε, ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη ΕΤΑ βεβαίω οι συνάδελφοι με τους οποίους είμαστε σε επαφή στον Καναδά φοβούνται το τι θα γίνει με τη ΣΕΤΑ, κυρίως για το τυρί. Γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ποσοστώσεις, ε, δεσμολογικές ποσοστώσεις ό,τι αφορά το τυρί. Και φοβούνται, γιατί εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει πίεση στο σύστημα των ποσοστώσεων και φοβούνται για το σύστημά τους. Όμως ε, μια αμφισβήτηση του συστήματος ε, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει αύξηση της παραγωγής ε, στον Καναδά και επομένως θα υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές. Και ένα μικρό σχόλιο. Αν συγκρίνεται στον Καναδά ουσιαστικά το κλάδο του βόλου είναι εντελώς απορριθμισμένος, το σύστημα το γαλακτοκομικό στον Καναδά έχει διατηρήσει τις ε, ποσοστώσεις. Τώρα, θα ήθελα κάτι να σας δείξω και θα ολοκληρώσω. Θα ήθελα να σας δείξω το χάρτη. Δεν ξέρω αν βλέπετε το χάρτη εδώ, με πράσινο. Έχουμε τις περιοχές που το 2014 είχαν την υψηλότερη παραγωγή γάλακτος ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στο διπλανό χάρτη με ροζ βλέπουμε τις περιοχές που κέρδισαν από την παραγωγή 2007-2014 και σε μπλε που έχασαν. Βλέπετε λοιπόν ότι το ίμιση των ευρωπαϊκών περιοχών έχασαν την περίοδο 2007-2014 και εκεί όπου είχαμε συγκέντρωση, ε, έχουν, αυτό ισχύει για τις περιοχές όπου είχαμε ήδη μεγάλη παραγωγή, τετραγωνικό χιλιόμετρο. Βλέπετε, κάτω χώρες υποχρεώθηκαν να θεσπίσουν ένα σύστημα περιορισμού ε, της ε, φόρτωσης των ζώων ε, σε γάλα, παραδείγματος χάρη, γιατί παρήγαγαν ολόνα και περισσότερο γάλα, αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν και την περιβαλλοντική οδηγία και επομένως δεν μπορούσαν να τη σεβαστούν. Έτσι λοιπόν έχουμε και ένα πρόβλημα από περιβαλλοντική σκοπιά που αφορά αυτή την γεωγραφική εξειδίκευση. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε εμείς. Συγχαρητήρια για τις απαντήσεις σας. Λυπάμαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητούμε όλα αυτά στο επισμένο χρόνο, όμως έχουμε ένα τελευταίο σημαντικό σημείο. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζω αμέσω με την ημερησία διάταξη και δι των υπαριθμών 6 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο οδηγίας, εκτελεστικής οδηγίας που τροποποιεί τα παρατήματα 1 έως 5 της οδηγίας 2029 σχετικά με μέτρα προστασίας κατά της εισόδου στην κοινότητα επιβλαβών οργανισμών και κατά της διάδοσής τους μέσα στο, στην επικράτεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την, τον νέο κανονισμό για τους επιβλαβείς οργανισμούς φυτών που παρουσιάστηκε στη διάρκεια του Οκτωβρίου στην Ολομέλεια δηλαδή του Στρασβούργου και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο επίσημο έντυπο. Η κυρία Αγγιλέρα που ε, κινείται από ιδιαίτερες ανησυχίες για τους επιλογές ορισμούς, όχι μόνο στην Ισπανία. Έχει εκφράσει τις ε, ε, ανησυχίες της αυτής στο σχέδιο οδηγίας. και για το σχετικό κανονισμό. Στην διάρκεια της τελευταίας συνάντησης της 8 Νοεμβρίου της Επιτροπής Γεωργίας παρουσιάστηκε το σχέδιο που υποβληθείτε στην Επιτροπή σήμερα θα κατεξαρθεί συμπληρωματική συζήτηση και πιθανώς πρώτα, ε, θα, ε, ψηφοφορία μάλλον της προτάσεως αύριο το πρωί για το σχέδιο του κ. Νταντέν. Και παρόντες είναι και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους υποβάλουμε σε λίγο. Προτείνω να λάβετε το λόγο λοιπόν στο τέλος μετά από τις παρεμβάσεις των ε, Ευρωβουλευτών και πρώτη η κυρία Αγγιλέρα για να εξηγήσει ε, την ε, πρότασή της. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα έχουμε και πάλι συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά είχα την αίσθηση ότι είχαμε ολοκληρώσει το, το θέμα στην προηγούμενη συζήτηση. Με περιπτώσει, η συζήτηση καλό κάνει στο μέτρο που διευκρινίζουμε πράγματα, γιατί όχι. Πρόκειται για ένα ψηφίσμα που αφορά το σχέδιο οδηγίας, εκτελεστικής οδηγίας, που τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 29 κάθετο 2000 για του τους οργανισμού οργανισμούς στα φυτά. Στις προηγούμενες συζητήσει είπαμε ότι θα έχουμε ένα νέο κανονισμό υγειονομική προστασία και θεωρώ ότι θα είναι καλό και όταν τεθεί σε ισχύ θα λύσει τα εκρεμή μας προβλήματα. Αυτό όμως το σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας αντιβαίνει σε κάποια εδάφια του κανονισμού που έχουμε εγκρίνει. Συγκεκριμένα, είναι ανεπαρκής ο φυτογειονομικός έλεγχος στα εσπεριδοειδή, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων. Δηλαδή, ανεπαρκής, επαναλαμβάνω, ο έλεγχος ο υγειονομικό έλεγχος που γίνεται στα εσπεριδοειδή ανάλογα με τον προορισμό τους. Δηλαδή, στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, όπως είπα, α, είναι, άλλος είναι ο έλεγχος αν προορίζονται για ε, κατανάλωση ως νοπαφρούτα ή αν προορίζονται για τη μεταποίηση. Ε, και έχουμε κυρίως ε, δύο επιβλαβείς οργανισμούς, ε, για τους οποίους ε, εντοπίσαμε ανεπαρκή φυτογειονομικό έλεγχο για τον καρκίνο των εσπεριδοειδών και την μαύρη κοιλίδα των εσπεριδοειδών. Είναι πολύ σημαντική επιβλαβής οργανισμοί για τα εσπεριδοειδή αυτά τα δύο, το citrus canker και η μαύρη κοιλίδα. Και δεν είναι θέμα συμφέροντος της Ισπανίας. Ε, το θέμα αυτό εξυπηρετεί την φυτοϊγειονομική κατάσταση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους επιβλαβείς οργανισμούς, ιδιαίτερα στα εσπεριδοειδή, αλλά είδαμε και τι έγινε με την ξυλέλα. Ε, και ε, την ξυλέλα ε, μας την έφερε στην Ευρώπη ένα, ένα φυτό καφέ. Δεν είναι ότι ήρθε από ένα ελαιόδεντρο και είδατε πώς έχει επεκταθεί στα ελαιόδεντρα της Ιταλίας η ξυλέλα. Δηλαδή, άσχετα με τον προορισμό των προϊόντων, η φυτογειονομική έλεγχη θα πρέπει να είναι επαρκής. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα νέο σύστημα ελέγχου ανεξάρτητα από τον προορισμό των φρούτων. Αν δηλαδή προορίζεται σε κατανάλωση νοπή ή σε, στη μεταποιητική βιομηχανία. Ένα άλλο θέμα. Για, τον τρίτο επιβλαβή οργανισμό τον ε, Λέο, Κοτρίτη αναφέρεται στην εκτελεστική οδηγία ότι χρειάζεται αποτελεσματική αντιμετώπιση. Δεν συμφωνώ, γιατί δεν αναφέρεται ποια είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση. Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών θέλουμε ε, να απαιτείται ε, θεραπεία εμψυχρό και να διευκρινίζεται το θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης για, για τον τρίτη επιβλαβή οργανισμό. Όλες ε, οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν και για την, τον τρίτο επιβλαβή οργανισμό, λέω κοτρέτα, την εμψυχρό ε, θεραπεία. Εμείς γιατί δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τέτοια θεραπεία σε ψήξη. Δεν μπορούμε να είμαστε ελαστικοί σε αυτά τα τρία σημεία. Δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί στους φυτογενομικούς ελέγχους. Άσχετα με τον προορισμό των προϊόντων, θα πρέπει η έλεγχη να είναι εξίσου αυστηρή. Αυτό είναι τα βασικά προβλήματα και τα σοβαρά προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Δεν, δίνουμε τη δεν δείχνουμε τη δέουσα επιμέλεια στην εισαγωγή των επιβλαβών οργανισμών και στην επιμόλυνση από, από άλλα προϊόντα. Και αυτό δεν είναι θέμα διεθνού εμπορίου, ούτε των εσπεριδοειδών, ούτε άλλων προϊόντων. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή και εμπροκειμένου την γεωργική παραγωγή εσπεριδοειδών, όπου και αν βρίσκεται. Και αν ήταν άλλο το προϊόν, πάλι το ίδιο θα λέγαμε, αν ήταν άλλη καλλιέργεια. Αυτά ευχαριστώ και ελπίζω αύριο να ψηφίσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε την κυρία Αγγιλέρα. Σαφέστατη η παρουσίαση. Το λόγο έχει η κυρία Μίλλαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας κρύψω ότι ε, έχω ορισμένα προβλήματα με αυτό το ψήφισμα. Πρόκειται για κανονισμό, πρόκειται για εκτελεστικό κανονισμό. που θα, ε, ε, θα τεθεί σε ισχύ το 2020 κατά πέσα πιθανότητα. Και προωθούμε εδώ ένα ψήφισμα για μια εκτελεστική νομοθετική πράξη. Διερωτώ με, είναι ε, δεσμευτικό αυτό. Εάν και ακόμα ψηφίσουμε σήμερα ή αύριο, είναι δεσμευτικό το ψήφισμα μας αυτό. Νομίζω πως όχι. Και άλλωστε τίθεται το θέμα ότι Βεβαίως εμπιστεύομαι την ΕΦΣΑ, τον οργανισμό ΕΦΣΑ, ότι όντω θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευθεί η εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε μια φάση στάθμισης διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες που δεν θέλουμε να επηρεάσουμε με προβάλλοντας εμπόδια βιδασμολογικό χαρακτήρα και γι' αυτό εγώ τάσσομαι μάλλον υπέρ της απορρίψεως του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Εσεί κύριε Ντές. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε και την αγαπητή συνάδελφο Αγγιλέρα για την υποβολή της εκθέσεως. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι δηλαδή εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβλαβείς οργανισμοί από τρίτες χώρε και ότι απαιτούνται μέτρα. Ε, αμφιταλαντεύομαι κάπως σε ό,τι αφορά την ε, στάση μου αύριο στην ψηφοφορία. Θεωρώ πάντως ότι πρέπει να ακουστεί και το Συμβούλιο. Και εγώ πάντως ε, έχω εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία του Συμβουλίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι αναγκαία ψήξη και άλλα ή αν χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ε, εμπιστεύομαι τους ειδικού. Δεν έχει καμία σχέση απολύτως με μέσας, κυρία συνάδελφε. Μιλούμε σήμερα για αυτό το θέμα. Αύριο θα γίνει πάλι ψηφοφορία. Εδώ και χρόνια ζω αυτές τις διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και μία εβδομάδα αργότερα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο τώρα μετά από το πέρας της συνεδριάσεως και μέχρι 7 η ώρα να γίνει εκπόνηση του καταλόγου ψηφοφοριών. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο χρειάζεται τέτοια πίεση χρόνου και αυτό δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε άσκηση κριτικής. Εγώ ασκώ κριτική μόνο στην διαδικασία και θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε αν ίσως μπορούμε να ψηφίσουμε ε, σε μία εβδομάδα. Ε, αυτή την επιθυμία εκφράζει και η συνάδελφος Σράιερ, η οποία δυστυχώς κολλείεται να είναι παρούσα σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Ράνς. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Αγγιλέρα και να υποστηρίξω το αίτημά της. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Παρόμοιο ζήσαμε και με την ξυλέλα φαστιδιώσα που δυστυχώς έφτασε και στην Ισπανία. Εμφανίστηκαν κρούσματα στις Βαλεαρίδες νήσους. Και τώρα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ενδημική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι ενδημική λοιπόν η ξυλέλα, γιατί δεν έχουμε αρκετούς, αρκετές ασπίδες προστασίας ώστε να αποκρούμε τέτοια χωροκατακτητικά ή τέτοιους επιβλαβείς οργανισμούς που ε, προκαλούν βλάβες στις καλλιέργειές μας. Και μάλιστα ε, χρησιμοποιούνται με φυτογενομικά προϊόντα, αλλά ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αποτελεσματικά προϊόντα για να αντιμετωπίσουμε την ξυλέλα και τις νέες δύο αρρώστιες που μας επισήμανε η κυρία Αγγιλέρα. Μάλιστα το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαλάρωσε τους ελέγχους για τα σπεριδοειδή σε περίπτωση προορίζοντας τη μεταποίηση. Ήταν μια απόφαση που ελήφθη μια συγκεκριμένη στιγμή που υποτίθεται ότι είχε προσωρινό χαρακτήρα και τώρα αυτό το προσωρινό θέλει να το μετατρέψει σε μόνιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη χαλάρωση των ελέγχων. Γι' αυτό στηρίζω την πρόταση κυρία Αγγιλέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έλαβε το μάτι την απόφαση, αλλά μεταξύ βρήκαμε και το ε, και περιπτώσεις ε, καρκίνου των εσπεριδοειδών και την ε, μελανή κοιλίδα των εσπεριδοειδών. Θα μας συμβεί το ίδιο που μας έτυχε και με την ξυλέλα. Είχε λάβει μια προσωρινή επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν ανεπαρκής αυτή η προσωρινή λύση γιατί βρέθηκαν κρούσματα και αλλού ξυλέλας και σε άλλα ελαιόδευρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε επουδενή να συμφωνήσουμε να μετατρέψει αυτή την προσωρινή λύση σε οριστική. Γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την παραγωγή σπεριδοειδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Στυκάστρου. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι ήδη έδωσαν τις εξηγήσει. Εγώ υποστηρίζω όσα υπόθηκαν από την κυρία Αγγιλέρα και από την ε, κυρία Ράνς Καρσία, αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι, κυρία Ντες. Το πρόβλημα, Άλμπερτ, είναι ότι δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Διαφορετικά ε, θα υπήρχε δυνατότητα να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Είναι τεχνικό το πρόβλημα και θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι κάναμε εξαιρετική δουλειά, πολύ κουραστική, αλλά με σημαντικά αποτελέσματα και είναι ο κανονισμός και όλοι θα θυμάστε την έκθεση McIntyre. Δυστυχώς αυτή η πράξη της Κομισιόν δεν πηγαίνει προς την κατεύθυνση του δικού μας κανονισμού. Δηλαδή, αντί ουσιαστικά ε, να αναλαμβάνει προληπτική δράση, φαίνεται να πηγαίνει σε αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλτερ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι εγώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες ε, που εξέφερε ο κύριος Ντέσος προς την διαδικασία και εγώ θα ήθελα περισσότερο χρόνο γιατί όλη αυτή η βιασύνη και να πω κάτι ακόμη γιατί θα καταψηφίσω. Καταρχήν πρέπει να επενθυμίσουμε ότι πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες ακόμη και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες χώρες όπου δεν μπορούμε να παράγουμε σπυριδοειδή. Επομένως εξαρτόμαστε ολοκληρωτικά από τις εισαγωγές. Εμείς ε, είμαστε πράγματι κατά του ψηφίσματος αυτού, γιατί δεν είναι δυνατόν να δεκτούμε κάποιες τέτοιες βιαστικές ε, δράσεις και τα υπόλοιπα κατά τα λοιπά έχουν αποκλειστεί. Πρέπει να πω λοιπόν ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι στο ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βίτεμα. Να ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Αγγιλέρα για την κατάρτιση του ψηφίσματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους επιζήμιους οργανισμούς που προέρχονται κυρίως από τις τρίτες χώρες. Πρέπει να έχουμε ισχυρά μέτρα να το πετρέπουμε αυτό. Αλλά αν διαβάσω αυτή τη στιγμή αυτό το ψήφισμα, έχω μια κάποια αμφιβολία και μια ερώτηση. Γιατί μόνο για τα σπεριδοειδή να έχουμε ένα μέτρο και αυτό είναι η ψυχρή θεραπεία. Γιατί δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε και άλλα αποτελεσματικά μέτρα τα οποία να ληφθούν υπόψη και αν ε, λαμβάνεται μόνο υπόψη την ψυχρή θεραπεία τότε ουσιαστικά ε, περιορίζεστε μόνο σε αυτό, κάνετε τον εαυτό σας ευάλωτο και θα περιορίσετε την ε, νέα εισβολή, αλλά και κάποια μέτρα αποτελεσματικά που ίσως θα ήταν καλύτερα, θα αυξήσετε το κόστος και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη και το εξή. Καταρχήν, θα μπορούσε να έχει ένα αποτέλεσμα ε, προστατευτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τρίτες χώρες. Δεν ξέρω αν συμβατώ με τον ΠΟΕ και πράγματι αυτό θέλουμε ως Επιτροπή Γεωργίας. Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους επιβλαβείς οργανισμούς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά αν μόνο επικεντρώνεστε σε ψυχρή θεραπεία, ανησυχώ πάρα πολύ ότι είστε υπερβολικά προστατευτικοί και ότι θα ζημιώσετε το εμπόριο και θέλω να ζητήσω να το εξετάσετε περαιτέρω το θέμα και να αναβάλουμε την ψηφορία για την επόμενη Δευτέρα. Άκουσα από το ε, προσωπικό μου ότι μπορούμε να ψηφίσουμε την επόμενη Δευτέρα στην Άγκρη και όλα αυτά να προλάβουμε και να πάει και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ. να σας δώσω και την φιλανδική σκοπιά στη συζήτηση. Εμείς ε, εξαρτόμαστε λόγω του κλίματος και στη Φιλανδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες ε, εξαρτόμαστε από την εισαγωγή εσπεριδοειδών. Το συγκεκριμένο σχέδιο ψηφίσματος ε, θέλει να εμποδίσει την εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών, συμφωνώ, και από εμπορική άποψη δηλώνει ότι είναι ευθύνη των τρίτων χωρών να εξασφαλίσουν ότι οι εξαγωγές τους, ε, οι εξαγωγές προϊόντων τους ε, είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς. Δηλαδή ήδη υπάρχει μηχανισμός ε, που προβλέπει ότι σε περίπτωση που κάποια προϊόντα έχουν, φέρουν επιβλαβείς οργανισμούς θα επιβληθούν κυρώσεις. Γιατί λοιπόν να μην εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει τη συνεργασία και των ε, υγειονομικών ελεκτών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή μου υπενθυμίζει τη συζήτηση που είχαμε για τη βιολογική γεωργία και για τη ε, καλλιέργεια χωρίς ε, χώμα. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα από το αν κάποιος προέρχεται από το βορρά ή το νότο όλο και περισσότερο καταφθάνουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια κάποιοι οργανισμοί που ε, στη χώρα προέλευσής τους είναι ακίνδυνοι, αλλά δημιουργούν πρόβλημα σε περίπτωση που εισάγονται στη δική μας ε, επικράτεια. Είναι θέμα φυτογειονομικής προστασίας εδώ. Θυμηθείτε τι έγινε στη ζωική παραγωγή. Εκεί είχαμε την, το, πυρετό των βοηών που μα ήρθε από το βορρά, ενώ κανονικά έρχονταν από το νότο και κατέστρεψε ένα τμήμα του ζωικού κεφαλαίου τη βόρεια Ευρώπη. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη λοιπόν. Και αν η αλληλεγγύη αυτή εμφανίζεται σε μια προσωρινή αναβολή τη ψηφοφορία, καλώ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει την πυγμή και την αποφασιστικότητά του για να εξαλείψει τα φυτογειονομικά προβλήματα που μας έρχονται από άλλε περιοχές. Ευχαριστώ κύριε Ντάντα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Αντρέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είχαμε πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει τα μέτρα στις εισαγωγές. Έχουμε προσθέσει νέους ε, οργανισμούς, ε, το ματοτύμπιο και ενισχύσαμε τους ελέγχους για τους ε, υπάρχοντες επιβλαβείς οργανισμούς του καταλόγου, για το citrus canker, για τη μαύρη κοιλία των εσπεριδοειδών και την καρπόκαψα, citrus greening. Ενισχύσαμε τους ελέγχους και τα αυστηρά κριτήρια της εισαγωγής και δεν πιστεύουμε ότι αντιβαίνουμε στον νέο κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Απλώς προσθέτουμε αυστηρότερα μέτρα γιατί προσθέτουμε στον κατάλογο με τους επιβλαβείς οργανισμούς και νέους οργανισμούς. Και δεν νομίζω ότι κάνοντας πιο αυστηρούς ελέγχους αντιβαίνουμε ε, στον κανονισμό. Το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη μετατροπή σε χυμούς. Έχουμε κάποιους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς που εισάγουν καρπούς και είχαν ζητήσει διαφορετική μεταχείριση για τα πορτοκάλια που προορίζονται για μεταποίηση. Γι' αυτό και είχαμε την ε, νέα δίωδο εισαγωγή σε ένα κατεπήγον μέτρο για τα εσπεριδοειδή από την Ουρουγουάη, την Νότια Αφρική και την Βραζιλία. και πρόθεσή μας ήταν να, προσθέσουμε αυτό το νέο μέτρο οριζόντια στην νέα νομοθεσία, στον ισχύ για όλες τις χώρες και να μην προβλέπεται αυτή η δυνατότητα μόνο για τις τρεις συγκεκριμένε τρίτες χώρες. Τώρα, θεωρείτε ότι με την πρόταση αυτή αποδυναμώνεται η προστασία. Όχι. Αντίθετα. Και αν διαβάσετε την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Τροφίμων, θεωρεί και η ΕΦΣΑ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μεταχείριση αυτή και τη μεταπίεση. Και από τη στιγμή που κάποιο προϊόν εισάγεται και ε, παρακολουθείται και μάλιστα δεν είναι μολυσμένο με έναν επιβλαβή οργανισμό και ακολουθεί μια πλαισιωμένη διαδικασία, οριοθετημένη, η ΕΦΣΑ λέει από τη στιγμή που ε, σε, ε, έρχεται αυτό το προϊόν σε μια περιοχή που δεν έχει παραγωγές περιδοειδών, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό ακριβώ κάνουμε έχουμε συγκεκριμένο σημείο εισόδου, συγκεκριμένη παρακολούθηση των προϊόντων αυτών και λέμε ότι τα, απόβλητα θα πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα σε ζώνη που δεν υπάρχει φυτογειονομικός κίνδυνος. Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τη γνωμάτευση της ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Εμείς ε, στηριχθήκαμε στη γνώμη του ΕΠΟ για την περίπτωση αυτή, είτε για την καρπόκαψα, είτε για τον καρκίνο των εσπεριδοειδών. Και στην ε, αρμόδια επιτροπή έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Έχουμε δύο εδώ απόψεις. Η μία λέει να αφήσουμε τις τρίτες χώρες να αποφασίσουν ε, πώς θα αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τους επιβλαβείς οργανισμούς και βλέποντας και κάνοντας. Και υπάρχει και άλλη γνώμη που λέει ότι όταν γνωρίζουμε ότι μία θεραπεία είναι αποτελεσματική, γιατί να μην την αναφέρουμε ρητά και να αφήσουμε τις άλλες δυνατότητες αντιμετώπισης ε, ανοιχτέ. Ακόμη συνεχίζεται η συζήτηση στην Αρμόδια Επιτροπή. Μιλήστε για αυτή τη θεραπεία ψυχρό, τη θεραπεία σε ψήξη, ε, για φρούτα που φέρουν τον καρκίνο των σπεριδοειδών. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ε, η συζήτηση στην Επιτροπή. Τώρα για τη μεταποίηση, ούτε και εκεί έχουν ε, ολοκληρωθεί οι συζητήσει στην Επιτροπή, Πάντω ε, για τη μεταποίηση δεν βλέπουμε άλλη λύση. Γιατί είμαστε πλήρω ευθυγραμμισμένοι με την γνωμάτευση του ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων, και δεν βλέπουμε πώ θα μπορούσαμε να αλλάξουμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις στην ε, μόνιμη επιτροπή. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και τα σχόλιά σας και οι απόψεις σας ε, συζητώνται και στην Επιτροπή τη Μόνιμη γιατί ακούγονται οι διάφορες απόψεις των χωρών. Πάντως για τη μεταποίηση η μόνη λύση που προβλέπουμε είναι να διατηρηθεί αυτή η προσωρινή λύση και να δοθεί δυνατότητα και στι υπόλοιπε χώρε, υπό αυστηρού όρου όμω, που ευθυγραμμίζονται με την γνωμοδότηση του ΕΦΣΑ. Για τη θεραπεία συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για να δούμε αν θα βρούμε κάποια χρυσή τομή, κάποια μέση λύση που θα σέβεται με την τεχνολογική πρόοδο και θα λαμβάνει υπόψη και τις ε, πιθανές γνωστέ μεθόδους θεραπείας. Δεν έχουμε ακόμη αποκρισταλώσει τη γνώμη μας στην, ε, ούτε στη Μόνιμη Επιτροπή, ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτάθηκαν κάποιες λύσεις, ε, έγιναν συζητήσεις οι οποίες και συνεχίζονται. Οπότε, μετά την ενδεικτική ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή θα πρέπει να περάσει το θέμα και από το φίλτρο των τρίτων χωρών, γιατί θα γίνει κοινοποίηση στον ΠΟΗ και οι τρίτες χώρες έχουν δύο μήνες για να αντιδράσουν. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι το μέτρο το κρίνουμε εμείς κατάλληλο για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή επικράτεια, που θυγραμμίζεται με τα επιστημονικά πορίσματα και, και είναι ανάλογο και με το στόχο, παρόλα αυτά οι τρίτες χώρες έχουν μέσα σε 60 μέρες τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν. Να πούνε αν είναι δυνατόν, τα έχετε χάσει, να πούνε ναι, θα το συζητήσουμε υπάρχει και αυτό το φίλτρο των τρίτων χωρών. Θα πρέπει να έχουμε διαβούλευση και με τρίτες χώρε αφού θα περάσει αυτή η πρόταση από εμά. Και επαναλαμβάνω, αυτό θα γίνει μετά την ενδεικτική ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή με τα κράτη-μέλη. Αυτό ω προς τη διαδικασία. Σας είπα σε ποιο ε, στάδιο έχει φτάσει η συζήτηση. Πάντω επαναλαμβάνω, για τη μεταποίηση, για τα φρούτα που προορίζονται για μεταποίηση, δεν βλέπω που υπάρχει πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στο κείμενο όπως τα κατεπήγοντα μέτρα. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις διευκρινήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο διακύβευμα και θα πρέπει να υπάρχει γρήγορη παρέμβαση βάσει και των προτάσεων που ακούσαμε. Θα πρέπει να δούμε τι θα ψηφίσουμε αύριο. Η πρόταση ψηφίσματος ε, είναι σημαντική. Εγώ θα ήθελα να πω ότι τεχνικά ίσως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και τις 5 Δεκεμβρίου. Αυτή η προθεσμία επιτρέπει να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία ή θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Εγώ νομίζω ότι εδώ διακυβεύουμε ουσιαστικά το ψήφισμα που προτείνει η Κλάρα. Προκειμένου να έχει μια κάθετη και μια σταθερή θέση το Κοινοβούλιο. Ο Πάολο για να προσπαθώ να βρω μια λύση. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά στο να δοθεί κάποια αναστολή για κάποιες μέρες. Όμως η ανησυχία μου είναι αν θα προλάβουμε την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν είμαστε σίγουροι, να ρωτήσω τον Γραμματεία, ότι θα μπει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, δεν θα αλλάξει κάτι σε 4-5 μέρες, και παρόλα αυτά αμφιβάλλον θα μπορούν να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό που λέει η Γραμματεία, αν ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου. Εξακολουθούμε να μπορούμε να περάσουμε το ψήφισμα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Η Γραμματεία. Ναι, να προσθέσω κάτι. Υπολογίσαμε ότι τεχνικά είναι δυνατό να ψηφίσουμε στις 5 και να πάει στην Ολομέλεια, αλλά η από την προπόθεση ότι οι πολιτικές αρχές, δηλαδή η διάσκεψη των πρόεδρων που θα καταρτήσουν την ημερησία διάταξη, θα δεχτούν να μπει αυτή η ψηφοφορία στην ημερησία διάταξη της Ολομέλειας. Μπορούμε δηλαδή να καθυστερήσουμε μέχρι τις 5, αλλά πρέπει να μας υποστηρίξουν οι πολιτικές αρχές για να μπει στον προγραμματισμό τη Ολομέλειας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αφού είναι στην αυριανή συνεδρίαση να θέσουμε σε ψηφοφορία το κείμενο, γιατί διακυβεύονται πολλά και θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μία πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο.